Thank Κυρίες και κύριοι, σας χαίρομαι, ε, σας που μπορούμε σήμερα να οργανώσουμε την ακρόαση αυτή. Που έχουμε λοιπόν την ακρόαση αυτή ε, για τις χώρες της ε, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι ε, μπορούμε να καλωσορίσουμε τον ε, Γενικό ε, Γραμματέα για θέματα Νοτιοανατολικής Ασίας, τον κύριο Λίν, όπως βεβαίως και όλους τους άλλους ομιλητές. Καλωσορίζω όλους σας που ήρθατε σε αυτή την ακρόαση, η οποία μεταδίδεται και από το διαδίκτυο και είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι στα γραφεία τους παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που διαδραματίζονται στην αίθουσά μας. Χαίρομαι επίσης για το ότι αυτό σημαίνει ότι μας προσφέρει τη ευκαιρία να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε μία έκθεση που αφορά στο μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ε, ο κύριος Πίτε Κόχπερ που είναι παρόν. Δυστυχώς για μας έχει αναλάβει την έκθεση. Πρόεδρε, ε, διαμαρτύρομαι. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος, αποδεικτεί η διαμαρτυρία σας. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να υπογράψει συμφωνίες εταιρική σχέση με 7 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα οδηγήσει σε εμβάθυνση της συνεργασίας. Εξάλλου, οι σχέσεις αυτές με τις χώρες της ε, Νοτιοανατολικής Ασίας, οι σχέσεις αυτές είναι σημαντικές όχι μόνο για οικονομικούς και εμπορικούς ε, λόγους, αλλά τέτοιου είδους ε, συνεργασίες ε, δείχνουν ότι και πέρα από τα εμπορικά θέματα υπάρχουν άλλα τα οποία απασχολούν όλους μας, έχουν σημασία για την παγκόσμια πολιτική και την περιφερειακή πολιτική. Κατόπιν τούτου, επαναλαμβάνω, ε, οι σχέσεις είναι σημαντικές όχι μόνο για εμπορικούς λόγους. Όσο περισσότερο αλλάζει ο, λόγος, ο κόσμος, όσο περισσότερο διαπιστώνουμε ότι στην περιοχή εκεί ε, μετατοπίζονται ισορροπίες δυνάμεων και μάλιστα αυτό το εκμεταλλεύονται ορισμένες χώρες. Νομίζω τόσο σημαντικότερο είναι κατά την άποψή μου τουλάχιστον οι σχέσεις αυτές να εμβαθυντούν περισσότερο και να είμαστε κι εμείς περισσότερο σε θέση να συνδέσουμε τα συμφέροντά μας έτσι ώστε οι σχέσεις αυτές να αντέχουν και σε περιόδους κρίσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η ακρόση μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε όλα τα επίκαιρα θέματα από διάφορες οπτικές γωνίες. Έχουμε και άλλους συναντέλφους παρόντες, τον κύριο Βάρνεκε και άλλους ε, οι οποίοι θεωρώ ότι θα συμβάλλουν στο διάλογο για να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτές θέσεις και αυτό θα βοηθήσει και τον εισηγητή μας ε, και αυτός να προσφέρει ό,τι μπορεί καλύτερα. Καταρχήν λοιπόν θα λάβει το λόγο ο Γενικός Γραμματέας για να μας ενημερώσει για ε, την ε, ε, τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη Νότιο-Ανατολική Ασία και εμείς ε, θα εξετάσουμε το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι σχέσεις αυτές. Άλλοι ομιλητές θα ασχοληθούν με επιμέρους θέματα των σχέσεων αυτών και θα μας δείξουν, θα μας παρουσιάσουν το πώς μπορούμε να προβάλλουμε τις σχέσεις αυτές για να σημειωθεί πρόοδος. Θα έχουμε και μια ακαδημαϊκή εισήγηση που αφορά στην, ε, ε, στις εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Ασία. Πριν όμως προχωρήσουμε θα δώσω το λόγο στον ειδήμονα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα Ανατολικής Ασίας, τον κύριο Βέρνα Λάγκε. Κύριε Λάγκε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εξοχότατοι, αγαπητοί πρέσβεις, αγαπητέ ε, αναπληρωτή γενικέ γραμματέα σε ένα απλό μέλος, ε, το, για ένα απλό μέλος ε, που είναι πρόεδρος ε, της Επιτροπής αυτής, είναι πολύ σημαντικό το να αποσκαλείτε στη σημερινή συνάντηση. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ θερμότατα. Εμείς από την αντιπροσωπεία ΑΖΕΑΝ διατηρούμε τις σχέσεις μας με τις 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας από την πρώτη κιόλας μέρα που εξελέγει άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές, μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω και χαίρομαι πολύ που η Επιτροπή εξωτερικά. Εσωτερικών Υποθέσεων εξετάζει με μεγαλύτερη προσοχή την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες της περιοχής αλλά και για μας, τους Ευρωπαίους. Γιατί μέχρι τώρα ε, προκαλείται η εντύπωση ότι ο μεγάλος παίκτη ήταν η Κίνα και όχι τα 10 κράτη της ΑΖΕΑΝ. Κράτη τα οποία έχουν ένα μεγάλο οικονομικό δυναμικό έχουν διανύσει ένα μεγάλο δρόμο προς τη διαδικασία του εκδημοκρατισμού. Έχουν την αγκέντα της ΑΖΕΑΝ 2015 που μπορεί να μετατεθεί βέβαια το 2015 να γίνει 18 ή 19 αλλά έστω και έτσι μιλάμε για μια πολύ φιλόδοξη διαδικασία ολοκλήρωσης ε, στην περιοχή αυτή και χαίρομαι που έχουμε κοντά μας τον κύριο Ρόμπερτ Γκιόπελ, τον αντιπρόεδρο της ε, επιτροπή με τις χώρες ΑΖΕΑΝ. Είναι λοιπόν απόλυτα κατάλληλη η χρονική στιγμή για να εμβαθύνουμε στις ε, σχέσεις μας. Η ε, ΑΖΕΑΝ είναι, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την Ευρώπη, στρατηγική και πολιτική. Η ταχύτητα της διαδικασίας ολοκλήρωσης είναι εντυπωσιακή και η περιοχή ΑΖΕΑΝ που έχει αυτό το στόχο της ατζέντα του 2015, το είπα ήδη, ε, έχει συστήσει θεσμούς ε, που ενδιαφέρονται για σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι ευτυχές το γεγονός ότι έχουμε εδώ τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΑΖΕΑΝ από την Τζακάρτα. Οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω στην διαδικασία ειρήνευσης, τις εξελίξεις στην Ταϊλάνδη, τις διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη για να συζητήσουν εκκρεμή ε, ε, θέματα εδαφικής κυριαρχίας. Ε, υπάρχει η διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Πόμα, στην Μιανμάρ. Όλα αυτά είναι πολύ θετικές εξελίξεις. Επίσης και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώθηκε ουσιαστικά ουσιαστική πρόοδος. Έχει συσταθεί η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει εγκριθεί ένας χάρτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλές εξελίξεις στη σωστή κατεύθυνση. Ορισμένοι παρατηρητές και στο ανθρώπινο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, όλοι αυτοί οι παρατηρητές ε, χαιρετίζουν τις εξελίξεις, ίσως θα επιθυμούσαν μεγαλύτερη ταχύτητα. Βέβαια δεν πρέπει να πιέζουμε υπερβολικά τους εταίρους μας. Ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει η αρχή της μη ανάμιξης όπως επίσης και αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται με συνένεση. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι υπάρχει σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς όπου έχουμε αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και το νέο εργαλείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ένα εργαλείο με δυναμική και ε, εξέλιξη. Ε, ο πρόεδρος είπε ότι ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για την πρόοδο που έχει τεθεί με πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, Μαλαισία, Ταϊλάνδη μεταξύ αυτών και να κάνουμε τα πρώτα βήματα για να υπογραφεί και μια παρεμπερή συμφωνία με την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες. Και να πω και κάτι ανοιχτά που δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε το ότι η Κομισιόν είπε ότι δεν έχει ε, ε, προσωπικό για να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος. Μα πώς είναι δυνατόν, αν υπάρχει ένας τομέας όπου πρέπει να επιταχυνθεί η πρόοδος, επρόκειται ακριβώς για τις ε, συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών και εταιρικών σχέσεων. Άρα δηλαδή θα πρέπει να πιέσουμε για το θέμα του προσωπικού. Και θα ήταν πολύ καλύτερα αν μέσω πρόθεσμα μπορούσαμε να συστήσουμε μια Επιτροπή Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών με το σύνολο των χωρών ΑΣΕΑΝ. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Έτσι λοιπόν η έκθεση του κύριου Πιτικόφε ε, θα κατατεθεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα ε, βελτιώσει τις σχέσεις με την περιοχή προς όφελος και των δύο πλευρών. Και να προσθέσω και άλλα δύο σημεία που αφορούν στη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα κοινοβούλια των χωρών ΑΖΕΑΝ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια έχει συστήσει ε, περιφερειακές συνελεύσεις με τη Λατινική Αμερική, τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη, παράλληλα με τη συνέλευση των χωρών ΑΚΕ που μάλιστα συνεδριάζει σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Δυστυχώς με την ΑΖΕΑΝ έχουμε μια πιο χαλαρή σχέση, λιγότερο θεσμοθετημένη. Έχουμε την ε, συνάντηση κορυφής ε, Ευρώπης και των χωρών της περιοχής, ΑΖΕΜ. Και έχουμε και την ΑΖΕΠ, που έχει μια κοινοβουλευτική διάσταση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια είναι να εμβαθύνουμε στη σχέση αυτή. Και τώρα εξετάζεται κατά πόσον η επόμενη ΑΖΕΠ, δηλαδή η επόμενη κοινοβουλευτική εταιρική σχέση το 2014 θα οργανωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά κανόνα βέβαια αυτό γίνεται το Μάιο και ξέρετε του χρόνου το Μάιο έχουμε τις ευρωεκλογές. Εκτός λοιπόν από τους δύο αυτούς θεσμούς ΑΖΕΠ και ΑΖΕΜ είναι πολύ πολύ σημαντικό να ε, στηρίξουν περαιτέρω την ΆΙΠΑ, την Διακοινοβουλευτική Συνέλευση και να τη θεσμοθετήσουμε περαιτέρω. Και οι δύο αυτές διαδικασίες είναι συμπληρωματικές και μπορούν να ε, ενισχυθούν. Το ΑΖΕΑΜ είναι ένας, ε, μια κινητήρια δύναμη για την ολοκλήρωση ως εκ τούτου Θεωρώ ότι πρέπει να την στηρίξει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα με τις χώρες ΑΖΕΑΝ προς την κατεύθυνση της καλύτερης θεσμοθέτησης ε, των σχέσεων με τις χωρές ΑΖΕΑΝ στο σύνολό τους. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να συσταθεί μια συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών ΑΖΕΑΝ το πρότυπο άλλων συνελεύσεων που υπάρχουν ήδη. Και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν παράλληλα με τις συζητήσεις για ε, κοινά στοιχεία οι δύο αυτές περιοχές θα μπορούσαν στο, μέλλον να ενισχύσουν περαιτέρω την κοινοβουλευτική συνεργασία. Και ίσως αυτό το θέμα μπορεί να το συμπεριλάβει στην έκθεσή του κ. Πιτικόπφε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ευόντως των εργασιών της ακρόασης. Πρόεδρος, κύριε Λάγκεν, πάμε τώρα στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, τον απληρωτή Γενικού Γραμματέα του κυρίου Λίν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, αξιότιμε κύριε Μπροκ, αξιότιμε κύριε Ράγκα, πρόεδρε της Αντιπροσωπείας, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, εξοχότητες κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμού του Γενικού Γραμματέα της ΑΣΕΑΝ, του κ. Λιγλουμένου, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Θέλω επίσης να αποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να μεταφέρω και το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα προς όλους εσάς που είναι ότι οι χώρες ΑΣΕΑΝ δίνουν μεγάλη σημασία στις μακρόχρονες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να δίνουν τις προσπάθειές τους ώστε να συνεχίσουν οι σχέσεις αυτές από τις οποίες εποφελούνται και οι δύο πλευρές. Πριν συνεχίσω προς την εταιρική σχέση, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω κάποιες εξελίξεις κλειδί στην περιοχή. Οι κοινότητες της ΑΣΕΑΝ θα συνεχίσουν όπως έχουν επιταχυνθεί και τον τελευταίο καιρό οι προσπάθειες προς την ολοκλήρωση στην περιοχή. Πολλές από τις προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται σε όλους τους τομείς αξιών της κοινότητας ΑΣΕΑΝ. Υπάρχει πρόοδο σε θέματα πολιτικής ασφάλειας ή οικονομικής. Στο θέμα της ασφάλειας αναγνωρίζεται η συνθήκη του 1976, το PSC όπως ονομάζεται, και ο κώδικας διοντολογίας όσον αφορά τις σχέσεις στην περιοχή που αποτελούν τη βάση για την περιφερειακή ειρήνη για περισσότερες από 29 χώρες που είναι τα συμβαλόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Συμφωνία του Ιούλιο που μας πέρασε με το Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι το οποίο δείχνει την ε, επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, δέσμευσή της να συνεργαστεί. Η Αζέν είναι υπέρ του αφοπλισμού και της μης διάδοσης των ε, όπλων. Θέλει να είναι χωρίς πυρηνικά και η συνθήκη για την περιοχή χωρίς πυρηνικά όπλα υπογράφηκε από 10 χώρες προκειμένου να πετύχει το στόχο αυτό και συνεχίζει το διάλογο με χώρες που έχουν πυρηνικά προκειμένου να ενθαρρυνθούν να υπογράψουν το πρωτόκολλο της ε, Σανγκάη και η υπογραφή της δήλωσης της Σανγκάης πέρυσι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην αποστολή τη ΑΣΕΑΝ για να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε πλήρη εφαρμογή της δήλωσης. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξή μας. Η συνεργασία στα πλαίσια του Περιφερειακού Φόρουμ, του ΕΡΑ, και η Υπουργική Συνεδρίαση Υπουργών Άμυνας προχώρησαν καλά και περιλαμβάνουν πλέον πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες, ιδιαίτερα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το στοιχείο κλειδί προωθούμε τον διάλογο και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή ΑΣΕΑΝ, εντατικοποιεί τις προσπάθειές της, προκειμένου να τεθεί πλήρως εφαρμογή η δήλωση για την νότια θάλασσα της Κίνας και θέλουμε να υπάρξει αποτέλεσμα όσον αφορά τον κώδικα δεντολογίας για την περιοχή αυτή της νότιας θάλασσας της Κίνας. Όσον αφορά τώρα τις εξωτερικές σχέσεις, ο διάλογος της ΑΣΕΑΝ και η συνεργασία με τους εταίρους μας, η διαπεριφερειακή οργάνωση, αλλά και άλλες πλευρές, συνεχίζουν τις προσπάθειες και επεκτηνόμαστε. Είμαστε μια από τις πιο επιτυχείς περιφερειακές οργανώσεις και αποτελούμε κινητήριο δύναμη για την ευημερία την, ε, και την ειρήνη. Πάνω από 17 χώρες που δεν είναι στην ΑΣΕΑΝ, οι οργανώσεις έχουν στείλει πρέσβες στην Ασιαν και 27 ασιατικές χώρες έχουν ε, αντίστοιχα αντιπροσώπους στον υπονάπτυξη κόσμου. Εντατικοποιούμε τις προσπάθειες λοιπόν για προώθηση της συνεργασίας με εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΑΣΕΑΝ οικονομικός πυλώνας έχει εφαρμόσει 80% των μέτρων τα οποία προβλέπονται ήδη με τεράστια πρόοδο σε διάφορους τομείς. Με αποτελέσματα πολύ συγκεκριμένα όπως είναι η μη, τα μη θεσμολογικά τέλη, όπως είναι άλλες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον ή με την διακίνηση υπηρεσιών και κεφαλαίων διασυνοριακά. Το 2015 λοιπόν θα είμαστε σε στέρα θεμέλια. Η οικονομική συνεργασία τώρα άρχισε μεταξύ ασιατικών χωρών και έξι εταίρους της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, μεταξύ άλλων Νέα Ζηλανδία, και το 2015 θα έχει ολοκληρωθεί. Κάτι το οποίο θέτει τα θεμέλια προκειμένου η περιοχή αυτή να αποτελέσει hub για οικονομικές δραστηριότητες. με πάνω από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, με 17 3 εκατομμύρια ΕΠ και 40% του παγκοσμίου εμπορίου. Με τις οικονομικές αυτές εξελίξεις θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω την οικονομική κατάσταση της περιοχής. Υπάρχει, εφόσον υπάρχει ανάκαμψη στην παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει και η με μια ανάπτυξη 5,3 με 6%. Ενώ πέρυσι ήταν 5,1%. Η οικονομία της ΑΣΕΑΝ είναι πιο ανταγωνιστική, με παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, που θα συνεχίσει στα πλαίσια της ζήτησης διαπεριφερειακά. Είμαστε παράδειγμα για πολλές χώρες στην περιοχή Πρέπει να ξέρετε ότι οι ορισμένες ασιατικές οικονομίες νιώθουν τον αντίκτυπο των καλών αυτών επιδόσεών μας. Υπάρχει και μεγαλύτερη ολοκλήρωση στον οικονομικό τομέα μεταξύ των χωρών ε, ΑΣΕΑΝ. Η επιδείνωση σε παγκόσμιο επίπεδο θα πειράσει βέβαια και τις κεφαλαιογορές στην ΑΣΕΑΝ. με επιπτώσει και στην πραγματική οικονομία. Συνεπώ οι οικονομικές αγορές προς το παρόν θεωρούμε ότι τα πηγαίνουν καλά παρά τις, ε, την ταραγμένη κατάσταση αλλού, αλλά βέβαια ανησυχούμε και εμείς για τη συνέχεια. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιες θα είναι επιπτώσεις στη συνέχεια για μας. Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις όμως. Η εξωτερική ζήτηση, οι τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, οι ανισορροπίες, όλα αυτά είναι προκλήσεις και για μας. Η κατάσταση όμως είναι γενικά θετική, γιατί παρά την παγκόσμια βεβαιότητα, κάτι το οποίο μας αναγκάζει σε μετριοπάθεια, παρόλα αυτά η οικονομική κατάσταση της ΑΣΕΑΝ θα είναι ισχυρή, θα είναι δυνατή, καλή. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η βελτίωση σε πολλές χώρες, ε, σαν σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, βάζει την περιοχή σε καλύτερη θέση προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει την παγκόσμια κρίση. Μείναμε σε αρκετά ισχυρή και καλή κατάσταση από τότε που ξέσπασε η κρίση και ο τραπεζικός και οικονομικός τομέας. Έτσι, αντιστοκόμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είχαμε αντισταθεί πριν από 10 χρόνια. Υπάρχει πρόοδος όμως και στον κοινωνικό τομέα. Κάτι πολύ βασικό για να έχουμε μια περιοχή που να έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο. Έχουμε αντιμετωπίσει μεταδοτικές ασθένειες με μέτρα τα οποία έχουμε εφαρμόσει και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία που θα νοιάζεται για τον άνθρωπο, που θα τον ανακουφίζει. Και αυτό το αποδεικνύουμε μετά τις διάφορες καταστροφές που έχουν πλήσει την περιοχή. Με ένα κέντρο για ανθρωπιστική βοήθεια. Η ΑΣΕΝ μπαίνει σε μία μακροχρόνια στρατηγική για να βελτιώσει και τη θεσμική κατάσταση στην περιοχή και για να συνδέσει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Για να το πετύχουμε αυτό, επικεντρωνόμαστε κυρίως στην σύνδεση την πραγματική αλλά και την εικονική. Και όλα αυτά βασιζόμαστε και στον ιδιωτικό τομέα και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την ανάπτυξη τώρα, η ΑΣΕΑΝ συνεχίζει να επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ικανοτήτων στην Καμπόδια, στο Λαό, στη Μιαμάρ και στο Βιετνάμ. Επίσης συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε ένα master plan για την διασύνδεση με στήριξη από τον ιδιωτικό τομέα που στηρίζει με τη σειρά του τις υποδομές. Τα επιτεύγματα είναι πολλά. Στην 22η διάσκεψη τον Απρίλιο που μας πέρασε, οι ηγέτες αποφάσισαν να ενώσουν τις προσπάθειές τους εν ώψη του 2015 και να αρχίσουν να δουλεύουν και σε σχέδια για μετά το 2015 αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, εξοχότες κυρίες και κύριοι. Θέλω τώρα να αναφερθώ στην σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΕΣΕΑΝ όσον αφορά την ασφάλεια. Έχουμε 30 χρόνια κλίση τέτοιων σχέσεων μεταξύ μας και επί τη ευκαιρία εγκρίθηκε και η δήλωση της Νιρεβέργης για την εταιρική αυτή σχέση που θέτει μακροχρόνιους στόχους και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και οι δύο πλευρές προς την κατεύθυνση κοινών στόχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια έχει εμπλακεί στην περιοχή της ΑΣΕΑΝ μέσω της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλογών. Και αυτό για να διασφαλιστεί η ειρήνη μέσω διαλόγου και συνεργασίας. Οι τακτικές υπουργικές συνεδριάσεις και οι ετήσιες διασκέψεις μετά τις υπουργικές οδήγησαν σε πολύ καρποφόρες ανταλλαγές απόψεων και διάλογο για θέματα αμοιβαίων ενδιαφέροντος. Προκειμένου βάσει αυτό να καθοδηγηθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Το εμπόριο, το συνολικό, αυξήθηκε 12,6%. 248,8 δισεκατομμύρια το 2011 και αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με ε, εκείνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι εισαγωγές αυξήθηκαν 15,3%. 1,82 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Έχουμε φτάσει σε 18,2 δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των χώρων ΑΣΕΑΝ με τις μεγαλύτερες κοινωνικές επενδύσεις. Προκειμένου να υπάρχει ευκαιρία για διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα και παραπάνω ευκαιρίες για ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, είχαμε και τη διάσκεψη επιχειρηματιών, που από το 2011 οργανώνεται κάθε χρόνο. Εκεί προσελκύονται διάφοροι επιχειρηματίες από την περιοχή ολόκληρη. Όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εταίρο για τις χώρες ΑΣΕΑΝ τα τελευταία χρόνια και στηρίζει την ε, οικοδόμηση ικανοτήτων. Είναι μια βοήθεια που αντιστοιχεί ακριβώς τη βοήθεια που χρειαζόμαστε εμείς. Βάσει το RISE και στα πλαίσια του διαλόγου που έχουμε μεταξύ μας, που αποτελεί ένα πολύ καρποφόρο παράδειγμα γιατί οδηγεί σε καλή, καλό συντονισμό μεταξύ μας και στηρίζεται έτσι η ολοκλήρωση στην περιοχή και η οικοδόμηση ικανοτήτων. Εκ μέρους λοιπόν της ΑΣΕΑΝ θέλω να αποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες μας και την εκτίμησή μας για την στήριξή σας και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να είσαστε ένας εταίρος κλειδί για τις χώρες της ΑΣΕΑΝ προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή τους στόχους μας για την περιφερειακή συνεργασία. Ελπίζουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την ΑΣΕΑΝ και μετά το 2015. Όσον αφορά τώρα τη νέα γενιά συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΣΙΑΝ, θα μπορούσε να επικεντρωθεί στα εξή. Πρώτον, ενίσχυση της εταιρική σχέσης με πραγματική εφαρμογή του σχεδίου δράσης Μπαντάρ Seri Μπαγκαβάν που αφορά την περίοδο 2013-2017 και εγκρίθηκε τον Απρίλιο που μας πέρασε, που έχει ως στόχο να επικεντρωθεί περισσότερο στο περιφερειακό επίπεδο η συνεργασία μας σε τομείς όπως είναι ο οικονομικός, ο κοινωνικός, ο πολιτικός κλπ. Δεύτερον, να υπάρξει διαβούλευση και συνεργασία σε διάφορα πολυμερή φόρα, Ηνωμένα Έθνη και άλλα, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και στην ΙΣΑΜ για να ενισχυθεί το πολυμερές σύστημα. Τρίτον, συνεχής διάλογος και συντονισμός σε θέματα περιφερειακά. Ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΑΣΕΑΝ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και περιφερειακός ε, διάλογος στα πλαίσια του Ασιατικού Φόρου που θα έχει σαν αποτέλεσμα να προωθηθούν θέματα κοινού συμφέροντος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ασάν, υπέρ της ειρήνης, της ευημερίας, της σταθερότητας. Τέταρτον, συνέχιση διημερών σχέσεων, πιο πολύ αντί για την ενίσχυση των ε, περιφερειακών δεσμών στην περιοχή. Θέλουμε την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου βάσει των δεδομένων που έχουμε από την ε, τοπική κοινωνία. 5. Εφαρμογή του Master Plan για την ασιατική κοινότητα. Επ' αυτού η ΑΣΕΑΝ θέλει να πάρει μαθήματα από την ευρωπαϊκή εμπειρία και να ετοιμάσει τα κατάλληλα συστήματα επικοινωνίας και διασύνδεσης που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες εχμής. Έπειτα, συνεργασία και ανάπτυξη. Πρέπει να καθοριστούν εδώ τομεί συνεργασίας που να αντιστοιχούν στις ανάγκες ανάπτυξης των χωρών ΑΣΕΑΝ και θα οδηγήσουν στην οικοδόμηση ικανοτήτων. Τέλος, θέλω να σας πω ότι η ΑΣΕΑΝ έχει παίξει ένα ρόλο κλειδί και εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο κλειδί για την ευημερία, τη σταθερότητα και την ειρήνη, αλλά και την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της περιοχής. Αποτελούμε κινητήρια δύναμη επίσης για την οικονομική ανάπτυξη. Παρά τις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, η ΑΣΕΑΝ εξακολουθεί να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπει τις δυνατότητες που έχει και προσβλέπει σε ενισχυμένη συνεργασία ΑΣΕΑΝ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε σε μια πολύ σημαντική στιγμή της συνεργασίας αυτής, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη βούληση από εκείνους που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις κατέρωθεν. Χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση για να συνεχιστεί αυτή η εταιρική σχέση, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα κάνουν τα λόγια πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον δεύτερο αγορητή, τον κύριο Βαρνέικε, αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή της ε, Asian Ευρώπης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι φίλοι κυρίες και κύριοι. Αποτελεί τιμή αλλά και χαρά για μένα που σας απευθύνω το λόγο. Θα ήθελα να σας μιλήσω αρχικά για την οργάνωσή μου. Είναι ένας οργανισμός ε, ο οποίος ασχολείται με τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΖΕΑΝ. Πρόκειται για ένα φόρουμ συζητήσεων που αποτελείται από 15 μέλη από την Ασία και την Ευρώπη και 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συν 10 ε, ακόμα κράτη της Ασίας και της Ευρώπης. Προσπαθούμε λοιπόν να φέρουμε μαζί, να ενώσουμε ε, την Ευρώπη και τις χώρες ΑΖΕΑΝ στο πλαίσιο μιας ε, ανοιχτή συνεργασία. Θα ήθελα να τονίσω πως εδώ δεν θα μιλήσω το όνομα του οργανισμού για τον οποίο εργάζομαι, ως διακυβερνητική οργάνωση. Η οργάνωσή μας δεν ε, συμμετέχει στις πολιτικές συζητήσει και εξελίξεις. Θα ήθελα όμω να αναφερθώ σε κάποιες γενικές ιδέες που προέκυψαν από 14 χρόνια επαγγελματική εμπειρία και σχέσεις με την Ασία και την Νότια Ασία ιδιαίτερα και ελπίζω να ε, είναι χρήσιμες σε όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ασία, από ό,τι γνωρίζω, είναι οι πιο ολοκληρωμένες οργανώσεις παγκοσμίω, αλλά διαφέρουν σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό της, ε, το μέγεθος, ε, των πληθυσμό κλπ. Επίσης ε, υπάρχουν και άλλες μερικές διαφορές ανάμεσα στις δύο που αφορούν στις προθέσεις ε, για την σύσταση αυτών των περιφερειακών οργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστάθηκε λόγω ενός πολιτικού οράματος για την δημιουργία ειρήνης αλλά και ευημερία στην Ήπειρο. Η οικονομική συνεργασία είναι τα μέσα για την επίτευξη του πολιτικού στόχου. Η ε, ΑΖΕΑΝ από την άλλη πλευρά ακολουθεί κατά την άποψή μου πρωτίστως ε, ένα οικονομικό όρομα. Ε, η Ασία θέλει να οδηγηθεί στην ευημερία αλλά και στην ειρήνη. Η περιοχή η οικονομική συνεργασία είναι ο τελικός στόχος. Ε, Άζιαν ε, βασίζεται στην απόκτηση μεγαλύτερου οικονομικού βάρους και ισχύω σε μια Ασία η οποία έχει δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ινδία. Αυτή η οικονομική, αυτό το οικονομικό όραμα προτίθεται να επιτύχουν μέσω συνεργασίας ε, ανάμεσα στις κοινωνίες των κρατών μέλων της οργάνωσης. Θετικές επιπτώσεις ε, ε, θα υπάρχουν στην ε, σταθερότητα και την ειρήνη, κάτι το οποίο μπορεί να, να ισορροπήσει και την οικονομική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη. Εν όψη των προθεσμιών, των χρονικών προθεσμιών, η Άζια θέλει να επιτύχει το στιγμότερο αυτούς στόχου το 2015 πάντως, αυτό το οποίο θα επιτευχθεί να μην είναι αναγκαστικά η πλήρης ολοκλήρωση τη εσωτερικής αγορά, αλλά ε, μια ε, καταγραφή των όσων έχουν γίνει και των όσων απομένουν να γίνουν. Αλλά ούτως ή άλλως η Άζιαν είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη δύναμη και αξίζει να τύχει μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης ε, στην περιοχή η οποία είναι είναι πατρίδα για τους περισσότερους ε, μουσουλμάνους θα έλεγα, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την αυξανόμενη σημασία της Ανατολικής Ασίας και της Αζιάν και αυτό αντανακλάται από την πολιτική που εφαρμόζεται τελευταία χρόνια στην περιοχή της Νοτιολογικής Ασίας και ειδικά στην ε, Νοτιοανατολική Ασία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου όταν ε, ασχολούμεθα με την περιοχή. Ε, το εμπόριο ανάμεσά μας ε, βαίνει αυξανόμενο συνεχώς, αλλά θα πρέπει να υποθέσουμε ότι και οι άλλοι έχουν την ίδια αντίληψη, όχι πάντα τα ίδια συμφέροντα, αλλά και στις προτεραιότητες. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ζήτημα πολιτικής πολιτική η Άζια από οικονομικής, και αυτά είναι σημαντικά να συνδυαστούν για το μέλλον των δύο περιοχών. Αυτές οι διαφορές όμως που υπάρχουν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρανοήσεις και να οδηγηθούμε σε δύο μονολόγους ε, χωρίς ε, να πετύχουμε την επιθυμητή συνεργασία. Τώρα, για τις ε, προκαταλήψεις, τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι όταν κοιτάνε την Ασία ή τις χώρες Άζιαν. Το Ίδρυμά μας ε, εξετάζει και τις δύο πλευρές. Έγινε μια μελέτη τα, στο 2010 και το 2012 στις χώρες σχετικά με την ανάλυση της πολιτικής κατάστασης για τις οικονομίες κλπ. Οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται την Ασία ως τις αναδυόμενες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένες της Κίνας και της ε, Ινδίας φυσικά. Και φαίνεται πως στην Ευρώπη οι πολίτες ε, δεν γνωρίζουν τη δυναμική αυτής της περιφέρειας. Ε, πάνω από 3.000 ε, ε, εφημερίδες αναλύθηκαν ε, σχετικά με, ανέλησαν μόνο σχετικά με το τι συζητιέται στην Ευρώπη και το τι έχουν γράψει διάφορα άρθρα. Στο κοινό πραγματικά ε, θεωρεί ότι η ΑΖΕΑΝ βρίσκεται κάτω από την ε, ναύτα σε ό,τι φορά τις ε, σχέσεις με την Ευρώπη. και κρίνουν πως η ΑΖΕΑΝ δεν αποτελεί προτεραιότητα. Φυσικά η ΑΖΕΑΝ έχει πολλή δουλειά μπροστά της να κάνει για να γνωρίζει, τα, να κάνει γνωστά το τι πράττει στην Ευρώπη. Έγινε μια μελέτη κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής κρίσης 53% ε, από τα 8.000 άρθρα που αναλύσαμε εξέρασαν ε, την οικονομική πτυχή αλλά κάποιες ε, θετικές οικονομικές ιστορίες πρόκειψαν κατά τη διάρκεια της περίοδου και ειδικά επιπτώσεις ε, της Ευρωζώνης στην ε, Νοτιοανατολική Ασία και η διασύνδεση ανάμεσα στις οικονομίες των Χροναζεάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική εταίρη μας ήταν φυσικά η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ε, Ασιάτες ερχόταν στην τρίτη θέση μετά από την Κίνα και την Ιαπωνία. Ε, λέξεις ε, όπως ε, αλαζονία ήταν αυτές που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο παράλληλα με την υποκρισία. Στην χώρα μου η κυρία Μέρκελ ήταν ο ηγέτης που αναφέρονταν περισσότερο στα άρθρα των εφημερίδων παράλληλα με τον Γάλλο Πρόεδρο αλλά και τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας ε, κ. Παπανδρέου. Οι χώρες Ασίας βλέπουν την Ευρώπη μόνο μέσω της ε, οικονομικής ισχύω. Ο κίνδυνος ε, Ευρώπη να γίνει ένας χώρος ε, δίδα την περάτα, διάρκεια βασίλειο δηλαδή, είναι σημαντικός. Και αυτό, αυτή η άποψη συμπληρώνεται από τις διάφορες προκαθορισμένες ιδέες και αντιλήψεις που υπάρχουν για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένωσης Άζιαν είναι, γίνονται όλο και πιο σημαντικές ε, και χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία και όχι ανταγωνισμός ε, ανάμεσα στα ε, δύο αυτές οργανώσεις. Πρέπει να προωθήσουμε το διάλογο με τον ASEAN συν δηλαδή των Άζιαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, τώρα το, ε, το πρόγραμμα Άζιαν συν 1 εμπεριέχει το κίνδυνο ότι μπορεί να ε, καθυστερήσει τις επιθυμητές για μας εξέλιξης. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να υπάρξει βελτίωση των ε, σχέσεων ε, και τα επιμέρους μέλη θα πρέπει να προωθήσουν και τις ε, διμερείς σχέσεις και να μην έρχονται σε ανταγωνισμό να υποκαταστήσουν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε λίγα από τα φόρουμ τα οποία οργανώνουν η Άζιαν με τις ΗΠΑ και φέτος για πρώτη φορά θα συμμετέχουμε στην ε, μη, ε, τυπικό, μη οργανωμένο διάλογο, μη τυπικό διάλογο που έδειξε στην Μανίλα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει συχνά ότι επιθυμεί να εμπλακεί όλο και περισσότερο με τις χώρες της Ασίας, αλλά θα πρέπει να καταστεί πιστικότερη στους χώρους και στα φόρα στα οποία συμμετέχει ήδη. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν σε τακτικές και σε υψηλό επίπεδο συναντήσεις. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα αυτό και ο διάλογος ε, με τις ΗΠΑ ξεκίνησε με νέα μορφή το 2009 ε, την δήλωση που είχε κάνει ε, τότε ο πρόεδρος Ομπάμα. Και υπήρξε συμμετοχή του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ στον επόμενο διάλογο. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη παρουσίας με το παράδειγμα της αμοιβαίας παρανόησης και να αναφερθώ στον στην σύνοδο του Νοεμβρίου 2007. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται περισσότερο με την ουσία και ε, έδειξε ότι η συνεδρίαση των προεξωτερικών εκείνης της χρονιάς που οδήγησε σε μια δήλωση ήταν ε, ιδιαίτερα συμβολική. Η Άτζαν πρόθεσε την ε, σύνοδο αυτή και όταν άνοιξαν οι θύρες ε, τη διασκεψής ε, αρχικά των κυβερνήσεων βρήκαν άνετες πολυθρόνες που τους ε, ανέμεναν. Ενώ οι μετέχοντες αλλά όχι μέλη κάθισαν σε κανονικές καρέκλες. Γιατί το λέω αυτό, διότι οι οργανωτές της Αζεν είπαν θα πρέπει να αισθανθείτε κι εσείς όπως αισθανόμαστε εμείς, πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και αυτή ήταν, ε, ε, αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρανόησης. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν ε, μπαίνουν σε μια αίθουσα συνεδριάσεων, τότε βλέπουν σε ποια θέση θα πρέπει να καθίσουν. Και αυτό αντανακλά τη σημασία που τους αποδίδει κάποιος. Εάν λοιπόν, έχει υποθεί ότι θα συμμετέχουν αρχικά των κυβερνήσεων, αυτούς περιμένουν να δουν ανάμεσά τους. Και αυτό είναι ένα σημάδι σεβασμού. Αυτή είναι η νοοτροπία τους. Και για να καταλήξω από η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ειδωθεί από την Άσεν ως ένας ε, ισότιμος ε, εταίρος σε υψηλό επίπεδο. Όχι ως ε, δάσκαλος ε, ή κήρυκας, αλλά ως ένας μεγάλος και ισχυρός ισότιμος συνομιλητής θέλουμε να γίνουμε δεχτοί ως, ως τη ούτη, τότε θα πρέπει να, γίνουμε, να εμφανιστούμε όπως ένας, ενιαίος, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η άζεν είναι σοβαρός εταίρος, αλλά αυτό θα πρέπει να το αποδείξει σε όλες τις συναντήσεις και να παίζει με την πρώτη ομάδα της και όχι με τους αναπληρωματικούς. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Τώρα λοιπόν <clears throat> με την ιδιότητά μου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθώσεων θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, πρέσβη ε, του Μπουρνέντα Ρεσαλάμ και νυν Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. I don't wish to add uh, more to what the, uh, the previous speaker has uh, said about ASEAN-EU relations, but let me just... Κοιτάξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω και εγώ λίγα λόγια για τον Μπουρνέι ε, Νταρουσαλάμ, το οποίο προεδρεύει φέτος στην ASEAN. Εμείς ε, έχουμε τη δική μας ερμηνεία για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Προεδρία και τώρα λοιπόν έχουμε περάσει ε, κάποιες δοκιμασίες. Η μεγαλύτερη βέβαια θα είναι τον Οκτώβριο όταν θα φιλοξενήσουμε την 23η Σύνοδο της ΑΖΕΑΝ. Όπως και όλοι οι άλλοι οργανισμοί και σε εμά υπάρχει το θέμα Τη οργάνωση που αυτό είναι πολύ σημαντικό προφανώς και για την ΑΣΕΑΝ. Γι' αυτό λοιπόν αν δείτε λιγάκι την ομάδα που θα επιληφθεί αυτή τη συνάντηση φέτο, θα διαπιστώσετε ότι τονίζουμε ιδιαίτερα θέματα που είναι σημαντικά για τους πολίτες, για τους νέους, θέματα που άπτονται της καθημερινής μας ζωής, της κλιματικής αλλαγής, του αναπτυξιακού χάσματος και παρεμφερή. Αυτά λοιπόν ε, θα παρουσιάσει φέτος η ομάδα μας ε, που θα ασχοληθεί με τους πολίτες και το μέλλον μας. Εμείς ε, θα κάνουμε απολογισμό στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ε, προσπάθειες της ΑΖΕΑΝ έτσι ώστε να μπορέσουμε μέχρι το 2015 να επιτύχουμε τις ε, φιλοδοξίες μας. Φέτος παραλάβαμε από το Λάος και θα παραδώσουμε στη Μιανμάρ. Έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο και θα επιτρέψουμε αρκετό χρόνο για να έρθουμε σε διαβουλεύσεις με όλες τις χώρες ΑΖΕΑΝ αλλά και με τις εταίρους μας για να συζητήσουμε όλα τα θέματα, κυρίως τα δύσκολα. Όπως είπε και ο αναπληρωτής ε, γενικός γραμματέας, ε, ασχολούμεθα με τις εξωτερικές μας σχέσεις κατόπιν τούτου και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσβλέπουμε στο να γίνει και η Νορβηγία μέλος της οργάνωσής μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και άλλα δύο θέματα να αναφέρω κύριε Πρόεδρε. Το ένα είναι η παρουσία της είπα της ε, εκπροσώπου πέρυσι στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και φέτος και πάλι. Αυτό είναι μια μαρτυρία για το πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ΑΣΕΑΝ. Θα ξανάρθει φέτος, τον Ιούλιο την περιμένουμε. Και τέλος, Πρόεδρε, ελπίζουμε να μπορέσουμε να καλωσορίσουμε και τις τον κύριο Λάγκε και την αντιπροσωπεία του εφέτος ε, στη συνάντησή μας. Ε, θα έχει ολοκληρώσει φαντάζομαι τότε τις επισκέψεις στις 10 χώρες ΑΖΕΑΝ και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν ε, κατόπιν και άλλες επισκέψεις. Και εμεί ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπιτικόφερ, ο εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον κύριο Βάρνικε και θέλω να μου επιτρέψετε να υποβάλω ερωτήσεις και στους δύο μετέχοντες στο πάνελ. Κύριε ε, Γενικέ Γραμματέα, εσείς ε, μιλήσατε για την ΑΣΕΑΝ που στοχεύει στους ανθρώπους και τη σχέση που υπάρχουν ανάμεσα στους λαούς. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε λιγάκι κατά την άποψή σας αυτό το, αυτή η δυνατότητα οι σχέσεις ανάμεσα στους πολίτες των χωρών ΑΣΕΑΝ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς μπορούν να εξελιχθούν. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Βάρνεκεν δεν εξετάσατε σε βάθος το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προαγωγή των σχέσεων. Ίσως λοιπόν επιθυμείτε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με αυτό. Και, και προς τους δύο μιλητές θέλω να κάνω μία ερώτηση που ε, μου προέκυψε μετά την παρατήρηση του κυρίου ε, Λάγκε κατά την εναρκτήρια ομιλία του. Είπε ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι ή δυνατόν να υπάρξει μια κοινοβουλευτική συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρός ΑΣΕΑΝ. Πιστεύετε εσείς ότι αυτό αξίζει τον κόπο. Ποια είναι η άποψή σας. Ε, Παρακαλώ. Κύριε Γέγκλη. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και το Προεδρείο και τους ομιλητές για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Μου επιτρέπετε να μιλήσω γερμανικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αμάν αυτός ο Κινέζ. Okay. Vielen Dank für die Informationen, die Sie uns gegeben haben, die uns teilweise auch nachdenklich äh, Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ε, είναι πολύ σωστές και συμφωνώ μαζί σας, κύριε Γενική Γραμματέα, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πράγματι ε, δεν είχαμε στρέψει την προσοχή μας ε, στις χώρες ΑΖΕΑΝ, στο σύνολό τους βεβαίως. Και είναι επίσης ε, σωστό που είπατε ότι οι μεμονωμένες χώρες ΑΖΕΑΝ και αυτές ε, δεν είχαν στρέψει την προσοχή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαν στρέψει περισσότερο την προσοχή τους σε μεμονωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είναι σωστό και αυτή είναι η τρίτη μου ερώτηση το ότι και τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από το οικονομικά συμφέροντα που είναι σημαντικά για όλους μας και πρέπει να προβάλλονται, ε, πρέπει να ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, όχι με μονομένα κράτη-μέλη. Ε, βεβαίως ε, μας ε, απασχολούν και πρέπει να λαμβάνουν με υπόψη μας ε, και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηθικής φύσεως. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά τα θέματα, διαπιστώνουμε ότι παράλληλα ο στόχος είναι να συσταθεί ζώνη ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Κάτι που νομίζω ότι το θέλουν και οι δύο ομάδες. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Εσείς ε, τι περιμένετε από εμά, τι πρέπει να γίνει ακόμα για να επιτύχουμε αυτό το στόχο από το δικό σας πρίσμα αλλά και από το πρίσμα του κυρίου Βάρνακε που ε, σε πάρα πολλά σημεία ε, αναφέρατε περιορισμούς. Τι μπορεί λοιπόν κανείς να κάνει και τι είναι απαραίτητο να γίνει. Και ίσως ε, μπορούμε να εργαστούμε για μια βελτίωση των σχέσεων ε, και πού ε, μπορούμε να επιτύχουμε κάτι συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Και συμφωνώ με πολλές από τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Φανερκέ. Όπως και ο κύριος Μπούτι Κόφερετς, και εγώ θα ήθελα να ξέρω τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η γνώση. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη στην Ινδονησία τα τελευταία δέκα χρόνια. είναι η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στη περιοχή. Και πώς λοιπόν βλέπουμε εμείς το θέμα της δημοκρατίας εκεί και στην περιοχή. Έχουμε τη Μιαμάρ, για παράδειγμα. Βέβαια και πέρα από αυτό. Κάποιος, στη διάσκεψη που έγινε εδώ δίπλα για την Ινδονησία σήμερα το πρωί, κάποιος μίλησε για τη μεγάλη σημασία που έχει το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας που φτιάχνει η Ινδονησία σήμερα. Και αυτό θα οδηγήσει σε διαφορετικές αντιλήψεις. Έρχομαι τώρα στο ρόλο της ΑΣΕΑΝ ως κάποιον που προσφέρει ασφάλεια στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την καταπολέμηση της πειρατείας. Αν καταφέραμε να έχουμε επιτυχίες στην καταπολέμηση της πειρατείας είναι χάρη της διάσκεψης αυτής για τον νόμο της θάλασσας. Πώς όμως όλα αυτά μπορούν να επεκταθούν περισσότερο και έτσι να μπορέσουμε να χειριστούμε τις εντάσεις που υπάρχουν και στην περιοχή. Όχι μόνο στη νότια θάλασσα της Κίνας αλλά και στη βόρεια. Κάποιος από το Ινστιτούτο της Σιγκαπούρης μου είπε σήμερα ότι πρέπει να περιμένουμε και άλλα για τις σχέσεις Κίνας, Ιαπωνία, Ιαπωνίας, ότι εκεί θα έχουμε περισσότερες εντάσεις από ό,τι στην Νότια Κινέζικη θάλασσα. Η ΑΣΕΑΝ τι μπορεί να κάνει γι' αυτά. Ευχαριστώ. Προτού να δώσω το λόγο στον επόμενο αγορητή, θα ήθελα να καλωσορίσω δύο βουλευτές από τη Βερμανία. Τον κύριο Βιν Χο, μέλος της, Επιτροπής, και τον κύριο Μιν Χο μέλος της Γερουσίας και οι δύο βρίσκονται ανάμεσά μας για μια επίσκεψη μελέτης. Καλώς ορίσατε. Bene. Mm, prossimo oratore. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Γκέμπελς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ Θα έλεγα πως μου άρεσαν πολλά από τα σχόλια του έρθω από την οργάνωση Ασία Ευρώπη που δήλωσε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αποδίδουμε παρά πολύ λίγη προσοχή στις σχέσεις μας με τις χώρες ΑΖΕΑΝ που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι φυσική μας εταίροι στην Ασία. Φυσικά έχουμε πολύ καλές οικονομικές σχέσεις αλλά και η συζήτηση το απέδειξε εξάλλου. Αλλά όταν μιλάμε για οικονομία, βιαζόμαστε να θίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πρωταρχική σημασία, αλλά έχω την εντύπωση πως ε, κάνουμε δηλώσεις ε, δηλωτικές θα έλεγα, καλή τέλεσης ε, που εμάς μας ακούν αλλά για τους ε, συναδέλφους από την ΑΖΕΑΝ είναι λίγο υποκριτικές ε, ή και λίγο επιφανειακές όπως είπατε. Ε, μιλάω για αυτά τα κατεπίγορα ψηφίσματα που περνάνε την πέμπτη το απόγευμα στο Στρασβούργο. Συμμετέχω σε συναντήσεις με τις χώρες ΑΖΕΑΝ από το 1995 και θεωρώ ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει εξελιχθεί σημαντικά όπως ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην τροφή, στην εκπαίδευση, στην εργασία, όπου τη χάνουν ε, στήριξης και προσοχής αλλά και εγγύηση από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζουμε την ε, πίεση που ασκείται στις ε, χώρες ΑΖΕΑΝ και ένα παράδειγμα πριν από μερικά χρόνια η Μιαμάρ πρόκειται να αναλάβει την Προεδρία της ΑΖΕΑΝ ε, την της Προεδρία όπως συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε το κοινοβούλιο μίλησε για στρατιωτική δικτατορία στην χώρα αυτή και πολλές χώρες της ε, ΑΖΕΑΝ ε, με διακριτικό τρόπο, δίχως ε, διακηρύξεις και δηλώσεις, φρόντισαν η Μιαμάρ να παραιτηθεί της Προεδρίας της ΑΖΕΑΝ. Νομίζω ότι αποτελεί μια καλή απόδειξη αυτής της πίεσης που ασκείται και εκδηλώνεται ορισμένες φορές σε κάποιες περιφερειακές ε, διενέξεις και διαφορές όπου άλλα κράτη-μέλη της ΑΖΕΑΝ ε, ενεργούν για να αποφύγουν το χειρότερο. Και κάτι ακόμα για το σχέσεις με τους ε, συναδέλφους των χωρών ΑΖΕΑΝ. Είχα την τύχη να εκπροσωπήσω το Ευρωκοινοβούλιο στην Λάιμπα ε, ΛΑΙΠΑ είναι ένα κοινοβούλιο που ψάχνεται, που είναι πολύ πιο τυπολατρικό και δεν ε, διαφωνώ το να υπάρξει ε, μια προσπάθεια δημιουργίας ε, μια σχέση όπως αυτή με τις ΑΚΕ, με τις χώρες ΕΣΑΝ. Λέγεται ότι θα πρέπει να, υπάρξει διαρθρωμένος διάλογος με τους κοινοβουλευτικούς ε, εκπροσώπους που συναντώνται εν ιάψια στην ΛΑΙΠΑ. Πέρυσι ήμουνα παρόν όταν έγινε μια συζήτηση για την ε, διένεξη γύρω από την ε, θάλασσα της Νότιας Κίνας και εκεί είδαμε μια συζήτηση ιδιαίτερα ενθαρρυντική την οποία θα πρέπει να στηρίξουμε διότι πρόκειται για ένα ζήτημα υψηλή σημασίας για αυτήν την περιοχή του κόσμου και θα έχει επιπτώσεις επί του υπολείπου κόσμου, στην υπόλοιπη φίλη. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Έχετε το λόγο, κύριε Λίν, και μετά ο κύριος Μενάκια. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτησή σας σχετικά με την ε, σχέση μεταξύ των λαών και το πώς πρέπει κανείς ε, να έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο. Εγώ νομίζω ότι για πολύ καιρό η ΑΣΕΑΝ ήταν ε, η εθερήτω μια γραφειοκρατική οργάνωση χωρίς να γνωρίζει κατ' ουσίαν τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν οι ηγέτες μας το γνωρίζουν αυτό και σε κάθε συνάντηση κορυφής συναντούμε εκπροσώπους των ΜΚΟ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ε, έχουμε μαζί τους μια τακτική επαφή. Έτσι λοιπόν στην τελευταία συνάντηση οι πολιτικοί μας ηγέτες ε, ήξεραν ότι έπρεπε να δώσουν σημασία στις ε, προσωπικές σχέσεις. Αυτό λοιπόν έπρεπε να φανεί περισσότερο, ότι είχαν συνειδητοποιήσει το θέμα του ανθρώπου. Άρα δηλαδή μιλάμε για μια άσεα που επικεντρώνεται πλέον στον πολίτη και νομίζω ότι είμαστε ε, στη σωστή κατεύθυνση και αυτό το γνωρίζουν οι ηγέτες μας. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των πολιτών, των λαών, νομίζω ότι για να το πετύχουμε αυτό Πρέπει να βελτιώσουμε τις σχέσεις, ε, να είναι πιο εύκολο να ταξιδέψει κανείς, άρα να βελτιωθούν και οι υποδομές. Υπάρχει λοιπόν ένα master plan για την διασύνδεση. Ε, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ε, θέματα, κυρίως όσον αφορά στην βελτίωση των υποδομών ε, έχουμε απευθυνθεί σε τέρους μας να μας πούν αν μπορούν να μας βοηθήσουν. Και για την ε, ε, διασύνδεση των πολιτών των λαών της περιοχής νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει με το να τους πείσουμε να ταξιδεύουν περισσότερο και με ανταλλαγές σε επίπεδο νέων, πανεπιστημίων, να υπάρχουν προγράμματα ανταλλαγών. Παραδείγματο χάρη στην περιοχή μας. Πηγαίνουμε τακτικά στην Κίνα ή στην Ιαπωνία. Ε, οργανώνονται αυτές οι συναντήσεις ε, νέων. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες διαπροσωπικές επαφές στην περιοχή μας. Επίσης, ε, να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση στα σχολεία για την περιοχή μας. Έτσι οι άνθρωποι θα γνωριστούν καλύτερα και σε βάθος μάλλον για να ξέρουν τι ακριβώς είναι η Ευρώπη και τι είναι η ΑΣΕΑΝ. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας, είπατε ότι υπάρχουν διαφορετικά ίσως ε, συμφέροντα μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσω. Όσον αφορά την ζώνη ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών, ε, προς το παρόν ε, νομίζω υπάρχει κάποια συμφωνία που έχει υπογραφεί η περιφερειακή ζώνη ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή και ελπίζω ότι ε, θα συνεχιστεί από τη στιγμή που θα θεσμοθετηθούμε κι εμείς. Πάντως προς το παρόν ε, συνεχίζουμε ε, αλλά νομίζω ότι μετά το 2015 θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Με ρωτήσατε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ολοκλήρωση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ε, να ε, καθορίσουμε κάποιες προτεραιότητες, να δούμε τι ακριβώς μας ενδιαφέρει μέχρι το 2015. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα που χρειαζόμαστε την αλληλένδεση Έχουμε λοιπόν προγράμματα ε, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, σχέσεις με τις χώρες που σας ανέφερα. Αν δείτε λοιπόν τα προγράμματα θα διαπιστώσετε ότι είναι προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν και αυτή τη στιγμή είναι προγράμματα ε, προτεραιότητας. Μπορούν λοιπόν να μας ε, βοηθήσουν Έχουμε όλοι μας εμπειρία από θέματα ολοκλήρωσης και πώς μπορεί κανείς να ε, βελτιώσει. Σε τεχνολογικό επίπεδο νομίζω ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε και ε, βεβαίως ε, αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε μία ε, κοινότητα μέχρι το 2015, ε, να έχουμε θεσμοθετηθεί. Αυτή είναι η τομή που μπορούμε να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τώρα άλλες ερωτήσεις, Νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι θα το απαντήσει ο αδελφό μου. Το δεύτερο κομμάτι αφορά στο ότι η ΑΣΕΑΝ μπορεί να προσφέρει ασφάλεια. Ε, μιλήσατε νομίζω και για την πειρατεία και για τέτοιου τους προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι προσφέρουμε ε, πλατφόρμες ε, διάρκειας ε, αξιόλογες στην περιοχή μας έτσι ώστε να μπορούν οι χώρες να συναντηθούν. Ε, Παραδείγματος χάρη το Asian Forum είναι το μόνο φόρουμ όπου και τα έξι μέρη είναι αποτελούν ε, μία πλατφόρμα για να μπορούν να συναντηθούν και να συζητήσουν άτυπα. Αυτή τη στιγμή οι διακομματικές ε, σχέσεις ε, δεν συνεχίζονται. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα. Κατά τα άλλα, αυτά είχα να πω. Νομίζω υπάρχουν και άλλες ε, πλατφόρμες, δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Καλύτερα να σταματήσω εδώ και να ε, παρακαλέσω στον συνάδελφό μου να συνεχίσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στον κύριο Μπάτικοφ για τις ανταλλαγές μεταξύ Ασιαν και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε από το Ίδρυμα Ευρώπης Ασίας κάποιες εμπειρίες στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Εκεί έχουμε ανταλλαγές. Όχι ότι φέρνουμε τον κόσμο από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις ανταλλαγές, τη συνεργασία. Ανθρώπους που παίρνουν πολιτικές αποφάσεις, καλλιτέχνες, δεν λέω ότι τους μεταφέρουμε από τη μία ήπειρο στην άλλη, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να έχουν τέτοιες ανταλλαγές να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα μέσω δικτύων που φτιάχνουμε. Και σας παρακαλώ κοιτάξτε την ιστοσελίδα μας ACF.tg και εκεί θα δείτε πολλά που γίνονται στα πλαίσια αυτά. Όσον αφορά τώρα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ρωτήσατε τι ρόλο θα μπορούσατε να παίξετε εσείς στα πλαίσια της ΑΣΙΑΝ, σκέφτηκα βέβαια το ΑΕΠΑ, που είναι η διακοινοβουλευτική συνέλευση. Ο συνάδελφος είπε ότι ακολουθεί ευρωπαϊκές προδιαγραφέ. Κοιτάξτε, θα ήταν σημαντικό να συμμετέχετε. Η Γερμανία, για παράδειγμα, συμμετέχει με κάποιο πρόγραμμα. Η γραμματεία μπορεί να βοηθήσει όσους δουλεύουν στις επιτροπές για τη δημιουργία δικτύων κλπ. Πάντως το σημαντικό είναι να συμμετέχετε στο ΑΙΠΑ και να δείτε ποιε είναι οι ανάγκες τους. Όχι να πάτε έτσι δυναμικά να επιβάλλετε κάτι, Απλώς να ψάξετε να δείτε ποιες είναι οι ανάγκες και ανάλογα με αυτές να δείτε τι έχει να προσφέρει η Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της ασφάλειας, όπου συμμετέχει ΑΣΙΑΝ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμπεριλαμβάνεται. Καλό θα ήταν να, να δείτε τι συζητάνε, τι τους ενδιαφέρει, τι ομάδες εργασίας έχουν, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν και να δείτε η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα έχει να προσφέρει και να το προσφέρετε. αν πρέπει να, έχει, να υπάρχει συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ, ε, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, δεν είναι δικό μου θέμα, το αφήνω σε εσά εντελώς. Η κύριε Γέγκλα τώρα. Μιλήσατε για την οικονομική πτυχή, για τα ηθικά ζητήματα, τις προδιαγραφές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται, δεν πρέπει να κρύβεται τίποτα από αυτά όταν συνεργάζεστε με την ΑΣΕΑΝ, εγώ απλώ θα σύστηνα να πείτε τη γνώμη σας, τι πιστεύετε, τι είναι σημαντικό για σας, αλλά να ακούσετε κιόλα, να ακούσετε τι έχει να πει άλλη πλευρά, τι τους ενδιαφέρει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ακούσετε ποιες είναι οι δικές τους ανησυχίες, που είναι διαφορετικές από τις ευρωπαϊκές. Αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σχετικά προβλήματα. Λοιπόν, ναι, να πείτε ποιες είναι οι δικές σας οι θέσεις, αλλά να ακούσετε και τους άλλους και να δείτε που υπάρχει κοινό τόπος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για πάρα πολλά θέματα. Κύριε Αγκόμες, αναφερθήκατε στην ασφάλεια. Όντως μια από τις πιο επιτυχείς συνεργασίες ήταν η δράση άξο που συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ΑΣΕΑΝ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και σε κάποια άλλη περιοχή, σε κάποια άλλη περίπτωση. Αλλά που ακριβώς αυτό θα το δούνε βέβαια οι κυβερνήσεις. Τέλος. Για τον συνάδελφό σας που αναφέρθηκε στην πίεση των ομολόγων, peer pressure. Ναι, φυσικά και παίζει ρόλο, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε πρόκειται για τις ΗΠΑ είτε για τη Ρωσία. Ε, φυσικά, όταν υπάρχει πίεση και εμείς ε, μέσα στην Ευρώπη προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση, πιέζουμε προς τη μία κατεύθυνση προς την άλλη. Εννοείται και στις χώρες σας αν το ίδιο συμβαίνει. Συνεπώς, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κοιτάμε πάντα ποιοι είναι εκεί που νιώθουμε ότι βρίσκονται πιο κοντά σε εμά που θέλουμε να τους στηρίξουμε. Ρωτήστε τους λοιπόν τι στήριξη θα θέλατε, τι έχετε να ζητήσετε και μαζί να φτιάχνουμε μια ατζέντα και να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, δηλαδή μέσα από το διάλογο. Ελπίζω έτσι να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας τώρα και ερχόμαστε στους τρεις επόμενους ομιλητές. Ο κύριος Τζόναθαν Χόλσλαχ είναι πρώτα, ο οποίος είναι ερευνητή από το Ινστιτούτο ε, Σύγχρονων ε, Κινέζικων Σπουδών των Βρυξελών. Στη συνέχεια, Κλάρα Πορτέλα, καθηγητής πολιτικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Και ο τρίτος είναι ο καθηγητής Γιούργεν Ρούλαντ, από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ. Μελέτες Νοτιοανατολικής Ασίας. Παρακαλώ, ο πρώτος που έχει το λόγο είναι ο κύριος Χολσλαχ. Μήπως να αλλάξουμε τη σειρά για να μιλήσει πρώτα κυρία Πορτέλα. Γιατί εσείς ήρθατε από τη Σιγκαπούρη, θα ήταν ε, ντροπή να σας αφήσουμε να περιμένετε. Θα πρότεινα λοιπόν να ξεκινήσει η δόκτωρ Κλάρα Πορτέλα και μετά ευχαρίστω να συνεχίσω εγώ. Μια που έρχεται από τόσο μακριά. Ευχαριστώ πολύ για την ευγένειά σας. Αλλά προτιμώ να ακολουθήσουμε τη σειρά. Θα είμαι πολύ σύντομος. Στην αρχική μου παρουσίαση Ξεκίνησαμε συζήτηση, την συζήτηση για τα στρατηγικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες αυτές. Ε, επίσης κοιτάξαμε το πώς ε, αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον και θα μπορούσα λοιπόν να τα αφήσω αυτά τα σημεία και να κάνω κάποιες προτάσεις αναφορικά με την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης όπως μπορείτε να διαβάσετε και στην έκθεση ε, η οποία είναι διαθέσιμη στην αίθουσα. Το βασικό μου επιχείρημα είναι ότι θα πρέπει να ε, δυναμώσουμε τις σχέσεις μας με την Αζιάν Είναι μια ζωτική σημασία σε εταιρική σχέση. Και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ε, πολλοί τόνισαν πως η ίδια συνεργασία είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή και θα πρέπει να ευαθυνθούν οι σχέσεις και οι δεσμοί. Πολλοί μίλησαν για τα γεωπολιτικά συμφέροντα τα οποία ε, θα έχει η Ευρώπη ενδυναμώνοντας την ολοκλήρωση των χωρών ΑΖΕΑ. Στο έγγραφό μου αναφέρω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και όταν μιλάμε για προχωρημένη συνεργασία τότε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν χρειάζεται να προσπαθεί συνεχώς να διευρύνει την ε, εταιρική σχέση με την ASEAN, ούτε να δημιουργήσει περαιτέρω κύκλους ε, συνεργασίας, αλλά να εντοπίσει σαφώς ποια είναι τα συμφέροντα, ποια είναι τα ενδιαφέροντα και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μόχλευση ανάμεσά μας. Στο έγγραφο επίσης προτείνω καταρχήν να θέσουμε σαφείς προτεραιότητες όταν μιλάμε για την ασφάλεια, θα νομίζω πως ε, οι σχέση ανάμεσα στην Άζιαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Δεν νομίζω πως ε, είναι σκόπιμο ή και απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να καταστεί ένας ε, πρωταγωνιστής στο ζήτημα της ασφάλειας στην περιοχή αλλά θα μπορούσε η Άζα να βοηθήσει και να συμβάλλει στο να υπάρξει μια μεγαλύτερη ισορροπία και να βοηθήσουμε εμείς με τη σειρά μας να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όταν πρόκειται λοιπόν τώρα για την οικονομική συνεργασία, να φτάνουμε στην οικονομική συνεργασία, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αυτό που προσδοκάμε. Ναι, φυσικά και έχει σημασία να ενισχύσουμε αλλά και να διευρύνουμε τις δυνατότητες για οικονομικές ε, συναλλαγές, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και τις επιπτώσεις ε, που μπορεί να δημιουργηθούν στα πιο αδύναμα κράτη της ε, χωρών Άζιαν στην Επιτροπή Εμπορίου κατέδειξα ότι θα υπάρξουν σημαντικός αντίκτυπος για τις φτωχότερες χώρες της ΑΖΕΑΝ. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων με την ΑΖΕΑΝ, τότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι χρειάζεται μια πολύ λεπτή και προχωρημένη εμπορική πολιτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα αμοιβαίας ε, ενδιαφέροντας, νομίζω ότι η αστικοποίηση είναι ε, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, μια πολύ σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι χώρες ΑΖΕΑΝ και φυσικά έχει ιδιαίτερη σημασία πέραν των ε, προτεραιοτήτων απαιτείται συντονισμός ε, πρωτίστως Υπάρχει ευρύ πεδίο για την δράση της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Κατάλαβα ότι υπήρχε ιδιαίτερο προβληματισμός αναφορικά με τον ρόλο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης αντί να ε, προωθήσει μια δική της πολιτικής, νομίζω ότι η προστέμενη αξία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης θα είναι να ενισχύσει τον συντονισμό με τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους, τους ενδιαφερόμενους, προτού να προτείνει νέες πρωτοβουλίες. Δεύτερον, στην ε, υπουργική συνάντηση, νομίζω ότι η υπηρεσία εξωτικής δράσης ε, θα μπορούσε να κάνει περισσότερα, έτσι ώστε να φτυγραμμίσει ε, τις πολιτικές που ακολουθούν από τις φυγγύλες πρωτεύουσες. Κάτι ακόμα και έχουμε επανειλημμένε συζητήσει για το θέμα αυτό. Ναι, έχουμε σημαντικά προγράμματα όπω ε, το θέμα στήριξη ε, τη περιφερειακή πολιτική, ε, το master plan, το οποίο θέλουμε να συμβάλλουμε και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν υποσχεθεί να ενισχύσουν, να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω. Νομίζω ότι μπορούμε να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθεια για τον συντονισμό. Επίσης υπάρχουν προτάσεις που βρίσκονται στο έγγραφό μου και που αφορούν ε, την ασφάλεια, την προαγωγή των επενδύσεων και ούτω καθεξής. Αλλά επειδή ο χρόνο πιέζει θα τα επιδείξω αυτά τα θέματα και θα τονίσω για μια ακόμα φορά ότι για μένα το μυστικό, το κλειδί για την ενίσχυση των σχέσεων με την Άζια είναι αποτελεσματικότητα και να καταστούμε πιο αποτελεσματικοί και πιο επιχειρησιακή στο πλαίσιο της ατζέντα που έχουμε θέσει. Ευχαριστούμε που ήσασταν σύντομο. Η κυρία Κλάρα Πορτέλα έχει το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Η παρουσίασή μου εμφανίζεται στην οθόνη νομίζω, ε. οπότε θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε. Πρόθεσή μου είναι να σας παρουσιάσω τις εξελίξεις, μια που έχουμε περιορισμένο χρόνο, τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη μελλοντική συνεργασία ΑΣΕΑΝ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το ξεκίνημα. Αρχικά, η ΑΣΕΑΝ δεν ήταν ένα σχέδιο ολοκλήρωσης ξεκίνησε μια οικονομική ολοκλήρωση στην αρχή της δεκαετίας του 90. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ΑΣΕΑΝ είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, που διαφέρει εντελώς από αυτά που γνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηρίζεται, θα έλεγα, ο τρόπος λειτουργίας της από την τήρηση της, και το σεβασμό της κυριαρχίας, από τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν μέσω διαβούλευσης και συνένεσης και αποφεύγουν τη δημόσια κριτική των υπολείπων μελών. Η κύρια εξέλιξη στη λειτουργία του οργανισμού ήρθε το 2007 με την χάρτα ΣΕΑΝ που εμπνεύστηκε από την επιθυμία να αλλάξει ΑΣΕΑΝ και να γίνει ένας οργανισμός που βασίζεται περισσότερο σε κανόνες με νομική υπόσταση και έτσι δημιουργήθηκαν τρεις κοινότητες. Θα μιλήσω για αυτές σε λίγο. Παρά το γεγονός ότι η υπογραφή της χάρτας αυτής αποτελεί ακρογωνίο λίθο για την θεσμοποίηση του οργανισμού που μέχρι τότε ήταν χωρίς προηγούμενο, διατηρήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της ΑΣΕΑΝ και παραμένει χωρίς κοινοβουλευτική διάσταση, ακόμα και μετά την υπογραφή δηλαδή της χάρτας αυτής. Υπάρχει μια πολύ αδύναμη κοινοβουλευτική διάσταση. Όσον αφορά τις τρεις κοινότητες, έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην εφαρμογή τους. Είναι πολύ διαφορετικές βέβαια από αυτές που γνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία είναι η κοινωνικοπολιτιστική Έχουμε μετά εκείνη για την ασφάλεια και τέλος την οικονομική κοινότητα. Η οικονομική κοινότητα είναι εκείνη που έχει και τον μεγαλύτερο παραλληλισμό με αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον τον πρώτο πυλώνα της. Οι άλλες δύο κοινότητες, πρώτα δημιουργήθηκε ένα σώμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην κοινωνική και πολιτιστική κοινότητα. Το γεγονός ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ διαφόρων μελών της ίδιας της ΑΣΕΑΝ, αλλά δεν συμμετέχουν όλοι στη συνεργασία αυτή, αυτό είναι χαρακτηριστικό, αλλά το ίδιο βλέπουμε και στον τομέα των πολιτικών και της ασφάλειας. Την κοινότητα δηλαδή, την πολιτική και της ασφάλειας. Και εκεί υπάρχει συνεργασία στον τομέα καταπολέμησης της πειρατείας, για παράδειγμα, όπου συμμετέχουν πολλά μέλη ΑΣΕΑΝ. Αυτό που είναι σημαντικό με τις εξελίξεις αυτές είναι ότι ότι υπάρχει ιδέα της ενισχυμένης συνεργασίας που εδώ και τόσο καιρό συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά έχει βρει το δρόμο της και ισχύει σε κάθε τομέα συνεργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας αναφέρω τώρα ποιε είναι οι τρέχουσες προκλήσεις. Κατά το παρελθόν η ποικιλομορφία. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε πολιτισμική διαφορά μεταξύ των μελών, αλλά και οικονομικές διαφορές και αυτά χαρακτήριζαν τα μέλη της ε, ΑΣΕΑΝ. Υπήρχε λοιπόν συνεργασία στην ΑΣΕΑΝ, αλλά χωρίς απαραίτητα να υπάρχει πάντα πρόοδος, γιατί υπήρχε αστάθεια σε κάποια μέλη της. Τελικά οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες ΑΣΕΑΝ σήμερα είναι η διαφορά που υπάρχει στην οικονομική ανάπτυξη και την ε, πολιτική ισχύ της Κίνας, που είναι βέβαια πολύ ανώτερη από εκείνη των υπολίτων. Η Κίνα δηλαδή κυριαρχεί και έτσι διχάζει κάπως τις χώρες ΑΣΑΝ. Έπειτα υπάρχει και το προφίλ της Ινδονησίας που ενισχύεται και ορισμένοι παρατηρητές λένε σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος η ελίτη της Ινδονησίας να εμποδίσει τις εξελίξεις σε άλλους τομείς στην ΑΣΕΑΝ. Δεν θα σας αναφέρω τώρα τα περί εξωτερικών σχέσεων, απλώς θα σας πω ότι η ΑΣΕΑΝ είναι ένας ανοιχτός οργανισμός. Έχει συνεργασία για διάφορες εκδηλώσεις στην περιοχή και έχει καταφέρει επιτυχώς να αποτελέσει το κέντρο στην περιοχή. Έρχομαι στην τελευταία μου διαφάνεια. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με τον οργανισμό αυτό που είναι για την περιφερειακή ολοκλήρωση αλλά που διαφέρει τόσο πολύ ως οργανισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ασία... πρώτα απ' όλα μπορεί να διατηρήσει τον κεντρικό χαρακτήρα της ΑΣΕΑΝ. Είναι σημαντικό το πολυμερές στοιχείο να διατηρηθεί. Δεύτερον, η εμβληματική προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια προς τις χώρες ΑΣΕΑΝ ήταν πάντα εκείνη για την ολοκλήρωση. Ο ρόλος αυτός όμως δεν είναι τόσο χαρακτηριστικός πια όπως ήταν. Και αυτό γιατί υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες και άλλοι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ψάξει να βρει και εναλλακτικού τρόπους συνεργασίας με τις χώρες ΑΣΕΑΝ, για να κάνει τη διαφορά δηλαδή. Όσον αφορά λοιπόν την βοήθεια αυτή για την ολοκλήρωση, εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τη δυνατότητα να συμμετέχει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια επίλυσης συγκρούσεων ή προβλημάτων, όπως έγινε στη Μιαμάρ, για παράδειγμα, όπου βοήθησε σε μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παίξει και ενδιαφέροντα ρόλο διαμεσολαβητή, προκειμένου να καθησυχαστούν διάφορες εντάσεις στην περιοχή. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μοιραστεί την εμπειρία που έχει στον τομέα της επίλυσης διαφορών για θέματα εδαφικά. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε. Ο καθηγητής Γιούργεν Ρούλαντ τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, το Προεδρείο και αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Η οικονομική κρίση της ε, Ασίας ε, ε, έχει προκαλέσει πολλές μεταρρυθμίσεις και αυτό αναφέρθηκε ήδη. Έχουν προκύψει ε, στόχο όπως είναι μεταξύ αυτών να υπάρξει μια κοινότητα μέχρι το 2015 να υπάρχουν ε, πιο αποτελεσματικές οργανώσεις και επίσης ε, να υπάρχουν και οργανώσεις που να στοχεύουν περισσότερο στον άνθρωπο. Με όλα αυτά έγιναν και άλλες σημαντικές αλλαγές διότι ο χάρτης περιλαμβάνει ε, και την ε, καλή διακυβέρνηση ως ε, ένα σημαντικό στόχο έτσι λοιπόν ο χάρτης της ΑΣΕΑΝ αποτελεί ένα ορόσημο στην εξέλιξη του οργανισμού παρά την απογοήτευση ορισμένων παρατηρητών. Ε, υπόσχεται πλέον περισσότερα δικαιώματα για τον πολίτη. Είναι ένας ε, οργανισμός ε, που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μια σχετική επιτροπή όπως και μια επιτροπή για την προγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Και αναφέρθηκε ότι υπάρχει και μία ε, δήλωση της ΑΣΕΑΝ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί λοιπόν περιλαμβάνονται όλα τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα που περιλαμβάνονται και στην διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όμως και άλλων ε, κοινωνικών και πολιτιστικών. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Ε, υπάρχουν ε, κριτικές φωνές που ακούγονται ότι σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις υπάρχουν πάρα πολλά κενά πολλοί επικρίνουν το ότι τα δικαιώματα αυτά ε, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από άλλες ε, συνθήκες. Ε, Παραδείγματο χάρη για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να ξεχνάμε όλο το πολιτιστικό υπόβαθρο που υπάρχει και ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και υποτίθεται αυτά δικαιολογούν την περικοπή δικαιωμάτων. Εδώ λοιπόν σας επαναλαμβάνω ε, υπάρχουν ε, ε, κατάλοιπα του παρελθόντος που πολλοί που ασκούν κριτική λένε ότι για αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση περικόπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφορά προφανώς όλες τις γενιές. Όλα αυτά δεν είναι λάθος, μόνο που πολύ συχνά αναφέρεται ότι αυτές οι τρεις γενιές και επίσης και τα έγγραφα της ΑΣΕΑΝ ε, δίνουν μεγάλη σημασία στα συλλογικά δικαιώματα και προβάλλουν ε, την παράδοση που ισχύει στην ε, περιοχή. Αυτό λοιπόν πολύ σωστά δημιουργεί επιφυλάξεις ε, στις ΜΚΟ και σε άλλους που λένε ότι η ανθρωπιστική παράδοση απλά χρησιμοποιείται ως πρόφαση για την περιστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μερικοί λένε ότι η Διακυβερνητική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, προστατεύει ε, δικαιώματα μόνο εφόσον υπάρχουν και ουσιαστικά συμφέροντα, εφόσον δηλαδή λάβουν ε, διαμαρτυρίες από ΜΚΟ και από πολίτες και τότε γίνεται ο έλεγχος και επιβάλλονται και ποινές. Αυτά όμως δεν εντάσσονται στο φορέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και περιορίζονται όλα αυτά μόνο στο να καταβάλλονται προσπάθειες. Κάτι άλλο. Μερικοί λένε ότι γίνεται παραπομπή στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ε, στηρίζει την ε, εθνική κυριαρχία αλλά μπορεί να αντιφάσκει με την ευθύνη προστασίας, ε, κάτι που ξεπερνάει την, τις ανησυχίες για την εθνική κυριαρχία. Το τέταρτο. Στα έγγραφα αυτά πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει δεσμευτικός χαρακτήρας. Δεν μπορεί κανείς να καταφύγει στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει σχετικό δικαστήριο στις χώρες Αζιάν και δεν προβλέπονται και κυρώσεις για τα κράτη που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις ε, του, των περί δικαιωμάτων. Και το τελευταίο που αναφέρεται είναι ότι δεν συμμετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Οι ασκούντες κριτικοί λένε ότι ε, κάποια κάποια μεταρρυθμιστικά μέτρα είναι γραμμένα σε μία ε, συγκαλυμμένη μορφή. Θα μπορούσα εδώ να αναφερθώ ε, στις κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις, τους οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών. Πολλοί λένε ότι Αυτά θυμίζουν κάπως τα αυταρχικά καθεστώτα της ε, δεκαετίας του 60 μέχρι το 80 και δίνουν ε, λαβή σε συμμετοχικές ε, διαδικασίες που δεν έχουν όμως σχέση με τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων παρά μόνο συμμετοχή στην χρήση αυτών των φορέων ως ημάντες για να γίνουν πιο αγαπητοί αυτές οι πολιτικές τους πολίτες. Σε εθνικό επίπεδο οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών είναι εκείνε που καλούνται να εφαρμόσουν αυτά τα νέα μέτρα. Η ΑΖΕΑΝ είναι αμυγός ε, διακυβερνητικός φορέας, άρα δηλαδή ε, η ευθύνη εναπόκειται στα χέρια των ε, κυβερνήσεων για να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα. Δεν θέλω να αναφερθώ πολύ σε αυτό, διότι υπάρχουν ε, διαφορετικά στοιχεία στις διάφορες χώρες. Δεν είναι ομοιόμορφη η εικόνα. Και σε μία σύντομη βιβλία δεν μπορεί κανείς ε, να αποδώσει δικαιοσύνη σε όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να υποθούν. Τώρα, όσον αφορά στο ότι δεν υπογράφουν οι χώρες αυτές ε, την ε, διακήρυξη των ΗΠΑ περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 37% των συμβάσεων έχουν επικυρωθεί. Υπάρχουν συνταγματικές ρήτρε. Πολλές από αυτές ε, αναφέρουν και τα μεμονωμένα δικαιώματα, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, σε ορισμένες χώρες υπάρχουν και ρήτρε περί δημοκρατίας. Υπάρχουν και παραλήψεις όπως η ισότητα των δύο φύλων, η ελευθερία άσκησης ε, θρησκευτικών πεπιθήσεων και αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι πολύ συχνά τα συντάγματα ε, χρησιμοποιούν κάποιες ιδιατυπώσεις ε, του στυλ ε, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Αυτό όμως μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα των πολιτών μέσα από νομοθετικές διαδικασίες. Έχουμε βέβαια αρκετούς νόμους και νομοθετικές διατάξεις που έχουν αναθεωρηθεί ή πρόκειται να αναθεωρηθούν. Η δικαστική εξουσία δημιουργεί προβλήματα. Σε κάποιες από τις χώρες ΑΖΕΑΝ έχουν συσταθεί συνταγματικά δικαστήρια. Θα ήθελα να παραπέμψω κυρίως το ρόλο του συνταγματικού δικαστηρίου της Ινδονησίας. Οι παρατηρητές λένε ότι εκεί δεν υπάρχει διαφθορά και έχει αρκετά μεγάλη αυτονομία, κυρίως οποτεδήποτε θεσμοθετεί και αποφαίνεται. Οι αστυνομικέ δυνάμεις είναι πρόβλημα. Δεν έχουν επαρκές προσωπικό, οι αμοιβέ δεν είναι ικανοποιητικέ. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω αναφερόμενος με λίγα λόγια στο τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική που ακολουθεί απέναντι στις χώρες ΑΣΕΑΝ. Εγώ δεν στηρίζω τις παλαιότερες ε, πολιτικές, γιατί αυτές βασίστηκαν κυρίως ε, σε υλικά πρόστιμα. Οι χώρες αυτές ε, αναπτύσσονται ταχύτατα οικονομικά έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες με την Κίνα και με άλλες αναδυόμενες χώρες και άρα οι οικονομικές κυρώσεις δεν είναι τόσο σημαντικές. Περισσότερη σημασία θα είχε να θίξει κανείς ε, την ε, επιθυμία που έχουν να αναγνωριστούν διεθνώς. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που έχουν καταδείξει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο. Και αυτό σημαίνει ότι οι χώρες Αζιάν πρέπει να επιπλήττονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συμμετρικό όμως, όχι ασύμετρο τρόπο. Θα μπορούσα να πω και πολλά για, τα, για την κοινοβουλευτική διάσταση του θέματος, αλλά θα προχωρήσω ίσως στη συζήτηση. Ωραία. Ο χρόνος δυστυχώς ε, λείπει. Συγγνώμη που χρειάζεται να δείξω στερότητα. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο, Μενέντες Δελβάλε και Γκόμες. Ε, παρακαλώ περιοριστείτε σε δύο λεπτά έκαστος, ε, διότι τα συμπεράσματα θα πρέπει να συνεργάγει ο συνέρφος Μπούτι Κόβερ που έχει το δικαίωμα να το πράξει ως ηγητής. Μενέντες, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είχα, δύο ερωτήσεις μάλλον μία ερώτηση σε δύο κομμάτια. Θα ζητήσω λοιπόν σε κάποιον από τους παρόντες ε, να απαντήσει. Φανταστούμε ότι βρισκόμαστε στην Ευρώπη και την επόμενη μέρα από την επίσημη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του, Προέδρου και του Κινέζου. Στην Ευρώπη κάθε ερευνητής, πολιτικός ή δημοσιογράφος μπορεί να θέσει μια ερώτηση σαν την παρακάτω ποια είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την συνάντηση του Κινέζου Προέδρου και του Ομπάμα. Υπάρχει λοιπόν ένα είδος συνοχής μεταξύ μας και στην περίπτωση αυτή της ερώτησης θα μπορούσε κάποια από τις ασιατικές χώρες να θέσει μια παρόμοια ερώτηση, δηλαδή ποια είναι η αντίδραση της ΑΖΕΑΝ ή ποια είναι η αντίδραση της χύψη χώρας. Υπάρχει λοιπόν μια παρόμοια συνοχή των χωρών ΑΖΕΑΝ που να επιτρέπει να υπάρχει αυτή η διάδραση. Ξέρετε, στην Ευρώπη μπορούμε να ρωτήσουμε την Κομισιόν, το Συμβούλιο να αντιδράσουν. Τέλειωσα, Πρόεδρε. Μεταν Γκόμες. Γκόμες, ένα σχόλιο. Μετά από τις παρατηρήσεις του κυρίου Γκόμπελς και του κυρίου Βάνε και παρατηρήσεις επί των παρατηρήσεων νομίζω ότι η πίεση ομοτύπων, ομοτήμων λειτουργεί όπως είπε ο κύριος Ρούλεντ εάν υπάρχει και μια άλλη πίεση. Αυτό είναι κάτι που λειτουργεί από τι δύο πλευρέ. Θα θέλαμε να ασκηθεί περισσότερη πίεση από του απλουσιάδε φίλου. για θέματα που αφορούν την Ευρώπη και συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή την Ουγγαρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιε είναι οι συνέπειε τη οικονομική κρίση και τη ανικανότητά μα αντιμετώπιση τη. Τώρα, οι ερωτήσει. Στον Τζόναθαν είναι επαΐων σε θέματα ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί η Άζαν να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των διαφόρων εντάσεων που υπάρχουν στον τομέα της ασφάλειας, ιδιαίτερα στην ε, Νότιο Ιαπωνία ή Κορέα. Μπορεί να κάνει λοιπόν διαφορά η Αζάν. Και τέλος προς τον ε, καθηγητή Ρούλαντ. Μιλήσατε για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, τις επιπτώσεις της κρίσης ε, για την τις χώρες ΑΖΕΑΝ. Τώρα Έχουμε το G8, έχουμε το G20, υπήρξε η διάσκεψη του Pittsburgh για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος, για, τον, για τους φορολογικούς παραδείσους. Η ASEAN συνεργάζεται για αυτά τα θέματα. Είναι ζωτικής φύσης θέμα και αφορά την συνολική διακυβέρνηση. Ωραία. Πέντε λεπτά. Απαντήσεις ε, φλάσου διότι θα πρέπει να, κάνει, βγάλει συμπεράσματα και ο εισηγητής. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. σε εγώ λοιπόν την απάντηση να ακούσουμε. Θα ζητήσω από τους συναδέρφους να απαντήσουν αντί για μένα, μια που δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Η απάντηση είναι όχι, φοβάμαι. Έχουμε μελετήσει το θέμα και το ενδιαφέρον είναι ότι είναι δύσκολο να υπάρξει συνοχή μέσα σε τέτοια φόρουμ. Στην Κίνα, για παράδειγμα, το έχουμε δει με την τελευταία διάσκεψη στην Καμπότζη, μετά την Υπουργική του Ιουλίου, φάνηκε αυτό με ανακοίνωση που έγινε ότι υπήρξε μεγάλος βαθμός διαφα... Ε, δια... Ε, διαφωνίας παρά τις προσπάθειες που γίναν. Να απαντήσω κι εγώ σύντομα στην κυρία Γκόμες. Ναι, η ΑΣΕΑΝ είναι σημαντικός παίκτη για την ασφάλεια στην περιοχή, ιδιαίτερα για την ε, νότια θάλασσα της Κίνας. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Προσπαθεί να παραμείνει συνεπής στις απόψεις της αλλά δεν ξέρω πού θα καταλήξει τελικά, αν δηλαδή όντως θα φανεί ένας ισχυρός εταίρος ή θα υποκύψει. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει και η Αμερική εκεί και να μην μείνει απομονωμένη ΑΣΕΑΝ. Κύριε Μπουτικόφερ, για τα συμπεράσματα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας για τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπαν. Έχω να κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω πραγματικά ότι αν θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ δύο οντοτήτων, είναι αδιανόητο η μία πλευρά να θέλει να είναι ο δάσκαλος και να περιμένει η άλλη πλευρά να είναι ο μαθητής. Δεν μπορεί. Η σχέση πρέπει να είναι αμοιβαία, δηλαδή να έχουν να μάθουν και οι δύο ο ένας από τον άλλον. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις παρατηρήσεις του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα όσον αφορά τα πυρηνικά. Πιστεύω ότι είναι μια κοινή προσπάθεια που πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε στην Ήπειρό μας. Δεύτερον, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανεβάσει το παιχνίδι της απέναντι στην ΑΣΕΑΝ και την περιοχή. Αρχίζει να το κάνει. Το υπογραμμίζω. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά, όπως υπόθηκε, έχουμε στη συνάντηση της Λάγκλα πρώτης τάξεως ε, συμμετοχή από την πλευρά μας, το δείχνει αυτό. Συμφωνώ και με αυτούς που λένε ότι από την μια μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία, από την άλλη μεριά τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να υποκαταστούν αυτή την ε, συνεργασία, αλλά να τη συμπληρώνουν. Τρίτον, για τις σχέσεις που θα έχουν σαν κέντρο τον άνθρωπο. Εδώ κρατάω ότι αν θέλουμε μεγάλη συνοχή σε ένα σώμα, σε έναν οργανισμό αυτού του είδους όπως είναι η ΑΣΕΑΝ, τότε όντως η σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι στοιχείο κλειδί. Το έχουμε δει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά που υπάρχει ζήτημα για το κατά πόσο οι πολίτες στηρίζουν μια πρόταση, ένα σχέδιο, εκεί έχουμε δυσκολία. Συνεπώς, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους είναι στοιχείο κλειδί και βλέπω να υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να τις προωθήσουμε αυτές τις σχέσεις. Τέλος, για τον καθηγητή Ρούλαντ, την κυρία Πορτέλα και τον ε, κύριο Χόλσλαχ. Και οι τρεις εντόπισαν διαφορές, διαφορετικές δυνατότητες προτεραιοτήτων στις οποίες θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε. Νομίζω ότι πρέπει όλες αυτές να τις αξιολογήσουμε πριν καταλήξουμε στην οριστική έκθεση της Επιτροπής μας για τις μελλοντικές σχέσεις ΑΣΕΑΝ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άξιζε τον κόπο η ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και σας Πρόεδρε και τους προσκεκλημένους μας, ε, βέβαια και ιδιαίτερα τον αναπληρωτή διευθυντή. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ όλους για τις παρουσιάσεις σας. Τώρα, περνάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε τώρα την παρουσίαση των μελετών με θέμα η εμπλοκή των οργασώσεων σαλαφιστών και ουαχαμπιστών στην υποστήριξη και την προμήθεια όπλων σε ομάδες ανταρτών ανά τον κόσμο. Σαλαφίστες ουαχαμπιστές. Η οικονομική υποστήριξή τους σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά ιδρύματα. Συναδελφοί, ερχόμαστε στην παρουσίαση των δύο μελετών λοιπόν, είπαμε εμπλοκή των οργανώσεων σαλαφιστών και χαμπιστών, εν ώψη της ε, έκθεσης της κυρίας Γκόμες που θα γίνει εκ μέρους της Επιτροπής μας για την ε, εμπλοκή των οργανώσεων αυτών στη Βόρεια Η πρώτη λοιπόν είναι η εμπλοκή των οργανώσεων ελαφιστων οχαμπιστών στην υποστήριξη και την προμήθεια όπλων σε ομάδες ανταρτών ανά τον κόσμο. Η δεύτερη μελέτη έχει να κάνει με την εμπλοκή των ε, οργανώσεων ελαφιστών και οπεχιστών στην οικονομική υποστήριξη εκπαιδευτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών ιδρυμάτων. Το λόγο έχουν οι συντάκτες. Ο κύριος ε, Ράσιμοφ είναι ο πρώτος και δεύτερο είναι ο κύριος Μονικέ από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ασφαλής και Πληροφορών των Βρυξελών. Καλώς ήρθατε, οι δυο σας. Παρακαλώ. Ποιος θα είναι ο πρώτος. Ο κύριος Ρασιμόρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Messieurs, bonjour. Je Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου την έρευνα που κάναμε για την οικονομική υποστήριξη των Σαλαφιστών και των αναχαμπιστών στις ε, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και σκεφτικές οργανώσεις και ιδρύματα. Καταρχήν η ομάδα μας ξεκίνησε από την αρχή ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στους αλαφιστές και τους οαχαβιστές και θα πρέπει να περιορίσουμε το εύρος της έρευνας στο επίπεδο των σαλαφιστών. Μια πρώτη διάκριση πολύ σημαντική είναι το γεγονός ότι οι ΟΑΜΠΙΣΤΕΣ συνδέονται άμεσα με ένα καθεστώς, με ένα πολύ καθεστώς που ισχύει στην Σαουδική Αραβία και ο γαλαξίας των σαλαφιστών συχνά είναι ανεξάρτητη των πολιτικών κομμάτων ε, και είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο ρεύμα των σαλαφιστών το οποίο είναι άμεσα πολιτικά συνδεδεμένο και ε, το άλλο κομμάτι του που θέλει να εμπλακεί στην, με την πολιτική βία. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλουμε, θέλ, θελήσαμε να διακρίνουμε είναι η δυναμική αυτής της οικονομικής στήριξης των σαλαφιστών και ουχαμπιστών στις ε, θρησκευτικές, θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα, διαφοροποιώντας τις ε, χώρες ε, όπου η χρηματοδότηση είναι ενεργή. Επιλέξαμε την Βοσνία και την Αίγυπτο, την Ισία, που θεωρήσαμε ότι είναι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για την προσέγγισή μας, το Πακιστάν, διότι η χώρα είναι γειτονεύει μάλλον με το Αφγανιστάν και πήραμε και την περίπτωση της Ινδονησίας. Βρισκόμαστε ενώπιν μιας αναδιόμενης οικονομικής δύναμης και νομίζω ότι ο όρος αναδυόμενο δεν είναι πλέον απαραίτητος διότι είναι μια μεγάλη οικονομική ασιατική δύναμη. Ως λοιπόν, περίπτωση της Αιγύπτου <clears throat> διαπιστώσαμε πως ο σαλαφισμός πρόσφατα εισήλθε στην πολιτική σκηνή. Πάντως κέρδισε τις τελευταίες προεδρικές εκλογές και αυτό αποτέλεσε έκπληξη για τους περισσότερους παρατηρητές διότι τα ρεύματα των Σαλαφιστών έλαβαν 125 έδρες στο ε, την Αιγυπτιακή Βουλή και είναι οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές θα έλεγα του κόμματος των αδερφών μουσουλμάνων το βασικό κίνημα των Σελαφιστών ε, ιδρύθηκε το 1926 και ε, αρνεί να ασκήσει πολιτική, δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ σε εκλογές και ε, το δόγμα του πρότεινε στα μέλη του να ε, απομακρυνθούν από κάθε πολιτική δράση και αυτό με βάση ενός νέες αρχέ που βρίσκουμε στα κινήματα των Σαλαφιστών ότι η πολιτική μπορεί να διχάσει και στη δίπτωση της Αιγύπτου με την, ε, το διχασμό των πιστών και άρα θα πρέπει να ε, μην ακολουθήσουμε τον πολιτικό δρόμο. Και αυτή η τάση σε μια αιτία διψτών με μια ριζική αλλαγή στον Αιγυπτιακό Σαλαφισμό μετά από την θάνατο του Προέδρου Νάσερ και την αποτυχία του νασερισμού στον Αίγυπτο και την έλευση του Σαντάτ με το άνοιγμα προς τον δυτικό κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Ο Ανουάρ Σαντάτ και η Σαουδική Αραβία υπόγραψαν τότε για πρώτη φορά μια συμφωνία. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό διότι από τότε ε, θα υπάρξουν δύο ρεύματα. Ένα ρεύμα ε, Αιγυπτίων φοιτητών που αναχωρούν για να ε, στρατευτούν στον μουσουλμανισμό και την εκπαίδευση των, στον Σούνιτ στην κατηγορία των Σουνιτών και την αποδοχή ενός ιδιαίτερα αυστηρού μουσουλμανισμού όπως αυτός που ισχύει στην Σαουδική Αραβία θα επιστρέψουν στην Αίγυπτο και θα αποτελέσουν τους εκπροσώπους ε, των Σαουδικών Αρχών που ξεκινούν τη χρηματοδότηση των ε, θρησκευτικών σχολιών, των ιερατείων και κάποιες ε, κάποια τεμένη. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον μια καταστάσεω που είναι πολύ κοντά στην στρατηγική που εφαρμόζουν οι αδελφοί μου Ρουμάνοι, οι ανταγωνιστέ του δηλαδή, δηλαδή να στηριχθούν στο κοινωνικό δίκτυο το, προκειμένου να ε, εγκατασταθούν ε, πολιτικά. δεν έχουμε βρει κάποια ίχνη πολιτικής ανάλυσης, ε, π.χ. ένα χρόνο πριν από τις ε, προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο μετά από την Επανάσταση, ότι το κίνημα των Σαλαφιστών θα μπορούσε να καταστεί η πρώτη δύναμη της αντιπολίτευσης. σε ό,τι φορά την πολιτική γραμμή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είναι λίγο νωρίς για να το αξιολογήσουμε Θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να προβλέψουμε, να προγνώσουμε ποιες είναι οι συμμαχίες ή οι διενέξεις, οι διαμάχες που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στους αριθμού μουσουλμάνους μακροπρόθεσμα και τους σαλαφιστές. Προς το παρόν βλέπετε τις εξελίξεις ότι η τάση, ε, μάλλον η ψαλίδα ανοίγει υπέρ της αντιπολίτευσης, ε, Βλέπουμε λοιπόν ότι το κύμα των ε, συνεχίζεται και οι πόροι προέρχονται από την Σαουδική Αραβία που βρίσκονται σε ανταγωνισμό με το Κατάρ, το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στους αδελφούς μουσουλμάνους. Υπάρχει λοιπόν μια πολιτική διαμάχη ανάμεσα στο Κατάρ και την Σαουδική Αραβία, που παίζεται σε αιγυπτιακό έδαφος, ε, όπως συμβαίνει εξάλλου σε άλλη περίπτωση με τον ε, Συρία περίπτωση λοιπόν της Τινησίας τώρα. Βρισκόμαστε σε κάτι το οποίο μας ε, κάνει να σκεφτόμαστε την Αίγυπτο. Σε μια πρώτη φάση έχουμε μια απομάκρυνση των Σελαφιστών ε, ε, από το πρώην καθεστώς, από το παρούμενο καθεστώς των και υπάρχει κάτι ακόμα στην περιοχή ότι οι σαλαφίστες, ε, οι σαλαφίστες δεν είναι καθαρά πολιτικού, πολιτικής χρειάς, αλλά προσπαθούν ε, να επηρεάσουν την κατάσταση και να επιβληθούν στους αριθμούς μουσουλμάνους μέσω του κόμματος ΣΕΝΑΝΤΑ. Θα υπάρξει λοιπόν μια συμφωνία αρχής. Ο Μπενελή θα επιτρέψει την κυκλοφορία προς την Σαουδική Αραβία των εκπροσώπων των Σαλαφιστών στην Τινησία και θα δεθούμε στην ίδια περίπτωση που γνωρίσαμε στην Αίγυπτο, δηλαδή ότι θα υπάρξει επιστροφή ελεγμένη, αλλά επιστροφή των χρηματοδοτήσεων προς την Τινησία και εδώ βρίσκουμε τον ε, διαχωρισμό που υπάρχει στην Αγγής Ανατολή σαλαφίστες που ε, στηρίζονται από τους αγαπητές και τους αλφούς μουσουλμάνους ε, που λαμβάνουν την επωνυμία τους ανάλογα με τη χώρα στην οποία δρούν. Στην Τινησία όμως ε, τα οργανώσεις των σαλαφιστών βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τους αλφούς μουσουλμάνους και θα βρεθούν σε μια θέση πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο αδιάλακτη από αυτήν της Αιγύπτου και οι ε, διαδηλώσεις και οι καθημερινές εκτροπές που διαπιστώνουμε καθημερινά στην ε, την Ισία ξεκίνησε από τις ε, πολιτοφυλακές, των, του θανάτου πρόκειται για δημιουργήματα των σαλαφιστών και όχι των Νάντα εδώ λοιπόν υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των δύο αυτών ρευμάτων που επιτρέπει τουλάχιστον στην Τινησία μια ριζοσπαστικοποίηση των τάσεων των σαλαφιστών που στηρίζει η Σαουδική Αραβία. Στην Βοσνία βρισκόμαστε σε μια διαφορετική περίπτωση. Ο Αχαμπιστές ε, προσωπούν μια, πολύ μικρή μερίδα του πληθυσμού. Εκτιμάται σήμερα πως υπάρχουν 3.000 άτομα τα οποία έχουν προσχωρήσει στα οργανώσεις των Σαλαφιστών στην Πεσνία, στο, πλαίσιο, στο σύνολο 1,5 ε, εκατομμυρίου περίπου μουσουλμάνων. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια αποτυχία σε ό,τι φορά την ε, εγκατάσταση αυτού του κινήματος. Αυτή η εγκατάσταση, ε, ε, μάλλον αυτή η στρατηγική εγκατάσταση ε, ανέρχεται στην περίοδο του φιλίου πολέμου στη Ιουγκοσλαβία και αφορά στη χρηματοδότηση μια σειράς ε, χωρών ε, για επί πολιτοφυλακών που στήριζαν ε, τον να στήριξη στη διάρκεια του πολέμου, ιδιαίτερα δούσαν υπέρ της Σερβίας ε, εν μεταξύ γνωρίζουμε ότι το Ιράν ε, έδωσε χρήματα στους ε, Σουνίτες και η Σοδική Ραβία ότι, είπε ότι προσέξτε διότι εμείς θα χορηγήσουμε πολύ σημαντικά ποσά που ανέρχονται την τελευταία χρονιά σε 350 εκατομμύρια δολάρια χρήματα λοιπόν τα οποία χορηγήθηκαν άμεσα για την αγορά και προμήθεια όπλων. στην Ρωσία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ. Βασίστηκαν λοιπόν στον, χρησιμοποίησαν μάλλον τον ε, πόλεμο της ε, Ιούκοσλαβίας, της πρώην Ιούκοσλαβίας, ε, για να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν κάποια κινήματα. Και εδώ μιλάμε για την στρατηγική την οποία εφάρμοσαν αυτοί των τεμένων και της χρηματοδότησης των ε, σχολείων. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια αποτυχία των ε, της Σαουδικής Αραβίας Υπάρχουν κάποιοι δείκτες που είναι ανησυχητικοί, διότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει στην Βοσνία προσπάθειες ε, που γίνονται από κάποια κινήματα που χρηματοδοτεί η Σαουδική Αραβία από το 2005 και εδώ μιλάμε για χρηματοδότηση των τρομοκρατικών κινημάτων και οργανώσεων. Η κατάσταση λοιπόν περιπλέκεται σημαντικά, βλέπετε λοιπόν του Πακιστάν. Βρίσκουμε την δέσμευση που είχε αναλάβει κατά τον πρώτο πόλεμο στο Αφγανιστάν, δηλαδή με την εισβολή των Σοβιετικών το 1979. Δεν θα σας αναφέρω τώρα το ολοστορικό της περιοχής, αλλά βρεθήκαμε σε μια παρόμοια κατάσταση, δηλαδή χρηματοδοτήσεις από πλευράς Σαουδικής Αραβίας με την στήριξη του πακιστανικού κράτους αλλά και της ε, πακιστανικής ασφάλειας ε, με την ίδρυμα σχολιών αλλά και οργανώσεων ε, φιλανθρωπικών και βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή από αυτή που υπάρχει στην την Ισία, την Αίγυπτο, την Βοσνία διότι η δημοκρατία είναι καθημερινή. Υπάρχουν απειλέ προς τις ΣΥΙΤΕΣ ειδικά, αλλά γενικά προς τη μειότητα των Πακιστανών και στην περιοχή Παστούν, δηλαδή στο βόρειο τμήμα της χώρας και την περιοχή του Καράτσι. Αυτή τη φορά λοιπόν εκ νέου βρισκόμαστε ενώπιον του αυτού μοντέλου δημιουργούν μια αλυσίδα ε, φιλαθροπικών ιδρυμάτων και τζαμιών δρώντας ε, προς όφελος ε, των ε, δυνάμεων ασφαλείας και του βαθέως κράτους. Έρχομαι στην Ινδονησία. Εδώ η στήριξη των Ουαχαμπιστών σε κινήματα, τα οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πολύ παραδοσιακά, η σχολή Αλμπαλή για παράδειγμα που προέρχεται από τους Αλαφιστές, τι διαπιστώνουμε. Διαπιστώνουμε στο Πακιστάν για παράδειγμα ότι οι αρχές δέχτηκαν και για να είμαστε δημοκρατικοί πρέπει να το πούμε ότι δέχτηκαν όλα τα ρεύματα του Ισλάμ και τα πιο αυστηρά υπό τον όρο ότι δεν θα παρεμβαίνουν και δεν θα ανακατεύονται σε παράνομες δραστηριότητες. Διαπιστώνουμε όμως ότι απέτυχε αυτό. Ενώ λοιπόν η συνήθις προκατάληψη που υπάρχει απέναντι σε ένα παραδοσιακό κίνημα λέει ότι αυτό δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στους σύγχρονους καιρούς, οι σελαφιστές και άλλα αντίστοιχα κινήματα μας δείχνουν ότι είναι πολύ ελαστικοί και προσαρμόζονται σε πολιτικές που ανοίγουν την πόρτα στην έλευση τους. Άρα διαπιστώνουμε ότι έχουν επιτυχεί σε πολλές και διαφορετικές περιοχές. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά θα σας μιλήσει και ο Κλόντ μετά γι' αυτά. Και θα σταματήσω για να μην ξεπεράσω το χρόνο μου. Ωραία, πολύ ενδιαφέροντο όλα αυτά. Ο κύριος Μονικέ θα μας εξηγήσει τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ επέλεξα να μην μιλήσω για κάθε χώρα χωριστά όσον αφορά την οικονομική στήριξη των σαλαφιστών και χαμπιστών σε τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά να θέσω το ζήτημα στο σωστό του πλαίσιο. Τι είναι οι σαλαφιστές, από πού προέρχονται, πού βρίσκονται σήμερα και πού πάνε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε καλά, ότι το σύγχρονο κίνημα των σαλαφιστών που έχει τάσει στη βία, το έχουμε στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική από τη δεκαετία του 70. Απαντάτε στην Αίγυπτο κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80 με επιθέσεις που έγιναν σε υψηλό επίπεδο με στόχο τουρίστες και τη δολοφονία του Σαντάτ το 1981 στόχος αυτής της εξέγερσης, γιατί για εξέγερση μπορούμε να μιλήσουμε στην Αίγυπτο, μια που έγιναν δεκάδες επιθέσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, κύρια βέβαια στο Κάιρο, αλλά όχι μόνο. Εκεί λοιπόν διαπιστώνουμε ότι υπήρχε μια σαφή στρατηγική, μια στρατηγική κατά μέτωπο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση της Αιγύπτου, γιατί, γιατί οι σελαφιστές και άλλοι από τον αραβικό κόσμο πίστευαν ότι δεν είχε νομιμότητα η κυβέρνηση στην Αίγυπτο επειδή δεν εφάρμοζε τη Σαριά, επειδή δεν ανταποκρινόταν στο μοντέλο εκείνο που ήθελαν οι σελαφιστές. Και επειδή βέβαια η Αίγυπτος είχε και ένα άλλο αμάρτημα στα μάτια των σελαφιστών ήταν οι σχέσεις της με το Ισραήλ. Άρα λοιπόν έπρεπε να τιμωρηθεί η Αίγυπτος. Έπρεπε να τη γονατίσουν. Και πώς θα τη γονάτισαν? Με στρατιωτικά χτυπήματα στην αστυνομία, στο στρατό, κατά του Πρόεδρου βέβαια, αλλά βάζοντάς τα και με τον τουρισμό στη χώρα, που ήταν και κύρια πηγή εσόδων για την Αίγυπτο την εποχή εκείνη. Ο συλλαφισμός όμως στην Αίγυπτο ιτήθηκε πήγε στην Αλγερία. Και εκεί τι διαπιστώσαμε. πώς φτάνει στην Αλγερία ο σελαφισμός. Υπάρχει μια στρατηγική που θα την συναντήσουμε ξανά αργότερα. Φτάνει μέσω καθηγητών δασκάλων που στέλνει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, σαλαφιστές που θέλει να τους ξεφορτωθεί η Αίγυπτος, τους στέλνει λοιπόν στην Αλγερία για να διδάξουν αραβικά, στα πλαίσια δηλαδή του προγράμματος εξαραβισμού που είχε τότε η κυβέρνηση της Αλγερίας. Ενισχύεται λοιπόν το κίνημα στην Αλγερία με επιπτώσεις βέβαια πολύ πιο σοβαρές από ό,τι στην Αίγυπτο γιατί οδήγησε σε εξέγερση μετά από τις εκλογές τέλος της δεκαετίας του 80 τέλος πάντων οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο στην Αλγερία με 150-200.000 νεκρούς. Πριν τα γεγονότα στη Συρία που έχουμε σήμερα, αυτά της Αλγερίας ήταν τα χειρότερα από μια εξέγερση σαλαφιστών. Ιτήθηκαν όμως. Όχι όμως τόσο πολύ όσο στην Αίγυπτο, ίσως γιατί Τους βρίσκουμε και σε πολλές άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή. Μέχρι μια κρίσιμη καμπή στην ε, ιστορία των σαλαφιστών τη σύγχρονη είναι η επέμβαση των Σοβιετικών στο, στο Αφγανιστάν. Είναι πράγματα γνωστά αυτά. Πάντως η αντίσταση προσελκύει στο Αφγανιστάν δεκάδες χιλιάδες εθελοντές από το Πακιστάν, από την Συρική Αραβία, την Αλγερία, από την Ευρώπη επίσης πήγανε μερικοί και από τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ασία, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν υπό την αιγύδα διαφόρων οργανώσεων που συνδέονται με τον ένα τον άλλο τρόπο με τους σαλαφιστές. Ακόμα και αν δεν είναι σαλαφιστές, ήταν αντιστασιακοί κατά των Σοβιετικών και της παρουσίας τους εκεί. Έχουμε τον Ζαν Μπαναντέν επίσης, έχουμε την ε, Αλκαΐδα η οποία αρχίζει να δημιουργείται από το 87-89 με πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Οπότε η επέμβαση των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα αυτή της παρουσίας των σαλαφιστών στην περιοχή. Επικεφαλής του, της Αλκαΐντα επίσης εμφανίστηκε αυτός που είναι τώρα μετά το θάνατο του Μπιν υπήρχε ένας πολιτικός στόχος, ενοποίηση. Εδώ και χρόνια ή και δεκάδες χρόνια αγωνίζεστε κατά των τοπικών κυβερνήσεων που σας καταπίζουν και θέλετε να αντιστρέψετε, ενώ στις χώρες σας τελικά βρίσκεστε σε ήττα. Ε, ενωθείτε. Αυτό ήταν το μήνυμα πρώτον. Δεύτερον, στρατηγική. Σταματήστε να εξαντλήσετε σε τοπικές επιθέσεις, αλλά κοιτάξτε πιο μακριά Γι' αυτό και υπάρχει θεωρία του κοντινού εχθρού αλλά και του μακρινού εχθρού. Ο κοντινό εχθρό είναι η κυβέρνηση που ο κάθε σαλαφιστή θέλει να ανατρέψει τη χώρα του, αλλά δεν τα καταφέρνει γιατί είναι πιο δυνατή από αυτόν. Αλλά ο πιο μακρινό εχθρό είναι οι πιο μακρινέ χώρε, ευρωπαϊκέ, Ηνωμένε Πολιτείε, που στηρίζουν την κυβέρνησή του, που δίνουν όπλα, που εκπαιδεύουν το στρατό, που διπλωματικά έχουν καλέ σχέσει κλπ. Αν λοιπόν με τη στρατηγική αυτή κατά του μακρινού εχθρού καταφέρνω να δυσαρεστεί απαρκώς τις Ηνωμένες και την Ευρώπη ώστε να αποκιστρωθούν από τον αραβικό κόσμο, τότε βρίσκομαι τέτα με την κυβέρνησή μου και μπορώ πιο εύκολα να την ε, νικήσω. Επίσης, οι Σελεφιστές προσπαθούν ε, να προβληθούν περισσότερο με οικονομική στήριξη σε διάφορα δίκτυα και οργανώσεις που έτσι, σιγά σιγά υπάρχει ανταλλαγή προσωπικού, ιδεών. Ας πούμε, οι Αλγερινοί κάνουν επιθέσεις ε, στην ε, Αίγυπτο για λογαριασμό των Αιγυπτίων ή οι Αιγύπτιοι για το λογαριασμό άλλων. Υπάρχει ένα παράδειγμα που δεν είναι βέβαια παράδειγμα εξέγερσης από το 98 Το πρωτάθλημα το παγκόσμιο ποδοσφαίρου στη Γαλλία όπου οι με την επιρροή της ε, Αλκαϊντα Τότε είχαμε ό,τι έμενε από την Τζία της Αλγερία. Είχαμε βέβαια και το 95 επιθέσεις. Αλλά εκεί το 98, ακόμα και εδώ στις Βρυξέλλες, οργανώθηκαν επιθέσεις κατά του Παρισιού, που ευτυχώς χάρη στην υπηρεσία πληροφοριών τη γαλλική και την γαλλική αστυνομία τελικά αποτράπηκαν και δεν έγιναν. Ο Μπενάντεν λοιπόν έχει την προπαγάνδα, τη στρατηγική, την οικονομική στήριξη και έτσι φτάνουμε και στη τζιχάντ των σαλαφιστών που βγήκε από την απομόνωση και πέρασε στην παγκοσμιοποίηση. Αυτή ήταν η πρώτη τροποποίηση. Η δεύτερη τροποποίηση είναι μετά το Σεπτέμβριο του 2001 που εκεί κλιμακώθηκε η δράση των σαλαφιστών και έχουμε τις επιθέσεις του 2001 και την επέμβαση μετά στο Αφγανιστάν, την εξαφάνιση των διαφόρων επιμέρους πλευρών. Κάτι το οποίο ενίσχυσε ένα κίνημα που υπήρχε ήδη σε ορισμένες χώρες και που του δώσαμε την ονομασία franchising, ότι δηλαδή δεν έχουμε πια μόνο την Αλκαϊντα που εκπροσωπεί τους αλαφιστές, όχι, βασίζεται και σε επιτόπους οργανώσεις. Σήμερα έχουμε 12 με 14 κινήματα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης των Σαλαφιστών, Σαχέλ, Βόρεια Αφρική, ε, Σουδική Αραβία, Τζίμι Σαμί στην ε, Νότιο ασια Ασία. Κάπου 12-14 διαφορετικές οργανώσεις ως προς την τακτική τους και το μέγεθός τους. Και βέβαια πολλούς υποστηρικτές στην Ευρώπη και στις Πολιτείες. Αυτό το franchising όπως το ονόμασα βοήθησε να επιβιώσει η Αλκαϊντα. Γιατί από τον Οκτώβριο του 2001 η Αλκαϊντα είναι το κέντρο και γύρω από τον, από τον Μπιν Λάντεν οργανώνεται η δράση τους, αλλά σιγά σιγά αποδυναμώνονται. Μπορούν να χρηματοδοτήσουν αντάρτες ή να κάνουν επιθέσεις και σιγά σιγά φτάνουμε στο τρίτο στάδιο, γιατί θέλω να μου κάνετε και ερωτήσεις μετά που είναι η ατομίκευση της τζιχάντ. Οι επιμέρους δράσεις δηλαδή στα πλαίσια της τζιχάντ. Ο σελαφισμός βρίσκεται σε ένα σημαντικό σημείο της εξέλιξής του. Ή ε, θα διαλυθεί ή θα ενισχυθεί κυρίως στη Σαχέλ και στη Συρία. Ανάλογα με το πώς θα προχωρήσουν οι συγκρούσεις στο Σαχέλ και στη Συρία, ο σελαφισμός θα υποχωρήσει ή αντίθετα θα επεκταθεί παρετέρω, θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο και θα έχει πιθανώς τη δυνατότητα να δράσει και αλλού, εκτός από εκεί που δράει σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκόμες είναι η πρώτη που έχει ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Γκόμες. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ για τα όσα μας ρωτήσατε. Πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτον, και ο κύριος Ρασιμόρα, μίλησατε πολύ για την Σαουδική Αραβία. Υπάρχει χώρα, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν ιδιώτες, υπάρχουν ομάδες Ε, αρχές θρησκευτικέ. Ο πρέσβης είναι εδώ, θα τον ακούσουμε δίχως άλλο της ε, Σουηδικής Αραβίας. Ακούσαμε τα λόγια σας, αλλά πώς κάνετε τη διάκριση για το τι είναι τι. τα πράγματα έχουν αλλάξει ή δεν έχουν αλλάξει στη Σαουδική Αραβία. Γιατί και αυτή ήταν αντικείμενο τρομοκρατικών ενεργειών. Ο τελευταίος στόχος της Αλκαΐντα. Και μια άλλη ερώτηση. Για τη σημερινή μορφή, κυρία Μονικέ, που έχει το κίνημα στη Σαχέλ και στη Σοδική Αραβία. Στη Βόρεια Αφρική, Κιμποαχάμ, στη Νιγερία. Από ό,τι φαίνεται, έχουν ένα πρόγραμμα ανάλογα με τις φυλές. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά. Και ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πιστεύετε εμείς να βοηθήσουμε ώστε το κίνημα αυτό να μην ενισχυθεί, να μην προσελκύσει περισσότερο κόσμο εκεί όπου δυσδύει. Romero López. No. Η κυρία Ρομέρο Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Θέλω να ε, σας ευχαριστήσω. Σας περιμέναμε και εδώ πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί για αυτά τα ζητήματα. Η αλήθεια όμως είναι ότι η γενική ενημέρωση που μας κάνετε πρέπει να μας κάνει να προχωρήσουμε περισσότερο σε βάθος, όπως είπε και η Άννα γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτή η δράση φιλανθρωπική που γίνεται δεν πρέπει να μας κάνει να ψάξουμε ποιος βρίσκεται από πίσω. Είναι χώρες, είναι ιδιωτικές οργανώσεις, είναι ιδρύματα. Η χρηματοδότηση των διεθνών μας κάνει τελικά μερικές φορές να τα βάζουμε με πολιτικά κόμματα τα οποία είναι δημοκρατικά. Η Ευρώπη φυσικά και θέλει να βοηθήσει στην ανάπτυξη, αλλά με κάποιο έλεγχο, ενώ σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει έλεγχος της χρηματοδότησης, τελικά φτάνει στην τρομοκρατία. Πέρα λοιπόν από τα χρηματοδοτικά δίκτυα υπάρχει και άλλος τρόπος να φρενάρουμε αυτές τις καταστάσεις. Να ξέρουμε τι εκπαιδευτικά ιδρύματα χρηματοδοτούμε, τι άλλου είδου ιδρύματα. Πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο για να ξέρουμε τι γίνεται και να μπορούμε να έχουμε στενή συνεργασία και να βοηθάμε τις χώρες τις οποίες, με τις οποίες θέλουμε να έχουμε συνεργασία, αλλά να ξέρουμε τι είδους συνεργασία έχουμε. Και θέλω να μιλήσουμε και για τις γυναίκες. Γιατί ο υπερεθρικισμός ε, μπορεί να μην πηγαίνει κατά εμπορικών δικαίων ή άλλων, αλλά κατά των δικαιωμάτων των γυναικών. Πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά τι γίνεται με τις γυναίκες. Κύριε Γιαννάκου, έχει το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες για την πρωτοβουλία που είχε ε, ώστε να μας ε, επισκεφθούν οι δύο ειδικοί και εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά που σχετίζονται με μια πολιτική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Αναδείξατε το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας ε, στην υπόθεση αυτή. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία διατηρεί σχέσεις με όλες τις δυτικές χώρες, πάρα πολύ στενές, και φοβούμε ότι κανείς δεν φύγει το ζήτημα αυτό ε, σε οποιαδήποτε ζητήματα έχουν σχέση με το εμπόριο, με την οικονομία, με το πετρέλαιο, με όλα τα υπόλοιπα. Ε, υπάρχουν οι φήμες που κυκλοφορούν για τη Σαουδική Αραβία ότι χρηματοδοτεί τις ομάδες αυτές. Ε, είναι γνωστό ότι οι οργανωμένες ομάδες παρεμβαίνουν στην παιδεία κυρίως και στο φιλανθρωπικό έργο και όπως θα ξέρετε ίσως ε, η Αίγυπτος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε παραδώσει στην ουσία την παιδεία και την ανώτατη εκπαίδευση, κολέγια και πανεπιστήμια πλην ελαχίστων όλα είχαν παραδοθεί σε αδελφότητες μουσουλμάνων. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Ε, Μένοντας σε αυτό το σημείο, ε, θεωρείτε ότι μπορεί ε, η Ευρώπη στα ζητήματα που αφορούν στην εξωτερική της πολιτική και τη σχέση με αυτές τις χώρες να θέτει τα ζητήματα αυτά χωρίς να θεωρηθεί ότι παρεμβαίνει σε παραδόσεις διότι φοβούμε ότι στις χώρες αυτές προβάλλεται πάντοτε ο ισχυρισμός ότι δήθεν είναι παράδοση Δηλαδή η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι παράδοση, η τήρηση της σαρία είναι παράδοση και άλλα τέτοια. Πώς θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδείξει αυτά τα θέματα ως παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ. Nikolai Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση για τον Σαλαβισμό στην Ευρώπη, δεν το θίξατε το ζήτημα. Δεύτερον, το θέμα των Φιλιππινών, ποιο είναι το μέλλον της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και του μετόπου. Και τρίτον, αν το κύμα του Μασαντ θα οδηγήσει σε ειρήνευση και ποιο είναι το μέλλον του σαλαβισμού εκεί. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τζιπ έχει το λόγο. Ε, Πρόεδρε, αυτά τα θέματα έχουν σχέση με την ιστορία της Αλκάιντα και με την ιστορία του Οσάμα Μπιν Λάντεν που από τη Σαουδική Αραβία πήγε στη Σομαλία και μετά στο Αφγανιστάν. Και σας ερωτώ, η άποψή σας μεταξύ ε, ουαχαμπισμού και σαλαφισμού ποια είναι. Υπήρχαν αυτές οι σχέσεις και κατά το παρελθόν. Υπήρχαν στενές σχέσεις ανάμεσα στους ουαχαμπίτες και τους σαλαφιστές. Μισό λεπτό. Έχω και άλλη μια δεύτερη ερώτηση. Ναι, αλλά δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος για την απάντηση. Εντάξει, τότε να είστε γρήγορος. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, αφήστε το. Μπορείτε λοιπόν να απαντήσετε οι ομιλητές. Δυστυχώς δεν έχουμε πλέον χρόνο, παρατηρεί ο Πρόεδρος. Θα είμαι σύντομος, η ερώτηση της κυρίας Γκόμες ε, για την Σαουδική Αραβία πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η εκθέση μας ε, δεν ε, κατακρίνει και δεν καταγγέλει το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας ε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλές σειράξεις Υπάρχουν προβλήματα και στη Σαουδική και στο Κατάρ και στην Τουρκία. Μπορούμε λοιπόν ε, να θεωρήσουμε απόλυτα θεμητό κατά τη διάρκεια του πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία οι μαχητές ε, να ενισχυθούν. Μπορούμε να θεωρήσουμε θεμητό οι μαχητές που αντιστέκονται στο καθεστώς του κ. Άσαντ να τη χάνουν στήριξη τουλάχιστον από ένα κομμάτι της Ευρώπης. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι πως ε, υπήρξε τακτικά στις περιπτώσεις που εμείς μελετήσαμε η συμμετοχή ενός Ισλάμ που είναι απόλυτο μιλάμε για το Ισλάμ των Οχαμπιστών που ταξιδιώτες, ε, φοιτητές, άτομα τα οποία ε, μετέβησαν στην Σοδική Αραβία ήρθαν ε, εμποτισμένα με αυτό τον ε, μουσουλμανισμό των Ουαχαμπιστών και οι ε, τοπικές, οι μάλλον οργανώσεις και χώρες ε, παίζουν τον ρόλο τους και είναι λογικό να βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία να χρηματοδοτεί φιλανθρωπικά ιδρύματα, είτε πρόκειται για δημόσια ή ιδιωτικά. Τώρα θίγεται ένα σημαντικό ερώτημα όταν ε, το 2005 στην Βοσνία εντόπισαν στην, ε, ότι μια φιλανθρωπική οργάνωση στο Πακιστάν αργότερα χρηματοδοτήθηκε από την Ισοδική Αραβή και χρησιμοποίησε τους πόρους ε, για να ε, χρηματοδοτήσει τρομοκράτες, ε, δεν υπάρχουν ε, τέτοιες αποδείξεις, αλλά εν πάση όπως είπε και κάποιος από τους συμμετέχοντες, η Σαουδική Αραβία ήταν θύμα της τρομοκρατίας πρωτίστως. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκα αλλά οι υπηρεσίες προφοριών ε, διαπιστώνουν ότι υπάρχουν οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από ε, ιδιωτικέ ε, οργανώσεις ή δημόσιες και τα χρήματα από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις εκτρέπονται και χορηγούνται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει λοιπόν κατηγορία εδώ για το ΡΙΑΝΤ ότι χρηματοδοτεί τον τρομοκρατία σε ό,τι αφορά, διότι θα μοιραστούμε τις απαντήσεις και θα προσπαθήσω να τα πω γρήγορα, το μέλλον του σελαφισμού στην Συρία, ε, περίπτωση νίκης του καθεστώτος του Μπασουάρα Ελασάντ. Σήμερα είναι δύσκολο να φανταστούμε μια συντριπτική νίκη. Κάτι το οποίο σημαίνει σφαγή αυτό βλέπουμε δηλαδή για 80 και 90 χιλιάδες νεκροί δεν θα, δεν θα είναι τίποτα. Η, στην περίπτωση αυτή η σύραξη θα συνεχιστεί και ανάμεσα στους μαχητές ε, σαλαφίστες ε, είναι πολλοί οι πιστεύουν ότι θα πρέπει να σου να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό θέλουν διότι θα βρεθούν και θα βρεθούν έτσι σε μια κατάσταση η οποία θα είναι κατά του πάνω τον επικίνδυνη. Όλοι λοιπόν έχουμε επέμβει στα τεκτονόμενα στη Συρία, η Ρωσία έχει τη δική της θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δική τους, η Ευρώπη το αυτό, το ίδιο σημαίνει και με το κατάρτιση στη Δυτική Αραβία, ε, το Ισραήλ, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ε, δύσκολη και δεν μπορούμε να ε, επικρίνουμε κάποιους. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε από πού ε, που κυκλοφορούν. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε με το ποιο είναι ο πάροχος των χρηματοδοτήσεων αυτών. Νομίζω ότι τέλειωσα τα πέντε με λεπτά που μου είχατε δώσει πρόεδρε. Ο συνάδελφος θα λάβει το λόγο. Για να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση της κυρίας Γκόμες, πριν περάσω στην πρώτη. Η σχέση των δύο αυτών κινημάτων, η ΑΚΜΗ, είναι καθαρά σαλαφιστική οργάνωση που βασίζεται στην επιθυμία των σαλαφιστών να φτιάξει καλυφάτα κτλ. Η Μπουαράμ δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια από μεγάλες επιθέσεις, κυρίως κατά των χριστιανών στην ε, Νιγηρία. Οι επιθέσεις κατά των αρχών εκεί, μεγάλες φαγές. Αυτό που βλέπουμε μετά την γαλλική παρέμβαση στο, Λαμί, είναι, στο Μαλί είναι να υπάρχει μια προσέγγιση μεταξύ των δύο, ενώ ήταν διακριτές όμοιροι από επαλλήλους της ε, Σουέζ που τους ε, απήγαγε δηλαδή η Μπαμάρ ήταν άνθρωποι της Μπουκαράμ που το κάνανε αυτό καθαρά για εγκληματικού λόγους για να βγάλουν χρήματα, λίτρα τα πήραν, δεν τα πήραν, δεν ξέρω από την ομοιρία αυτή η Μπουκαράμ εξάλλου χωρίστηκε στη, σε μια οργάνωση που έχει μια πολιτική ατζέντα που είναι πιο κοντά στην ακμή. Τώρα θα δούμε αν θα υπάρξει προσέγγιση τελικά με την ακμή. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αυτά που γίνονται στο Σαχέλ μπορεί να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρη την περιοχή και τον Ήγερα και τη Μαυριτανία, αλλά και το Καμερούν, ακόμα ή την Ιγυρία. Για τον σελαφισμό στην Ευρώπη τώρα. 14 βιβλία και δύο ώρες συζήτηση θα άξιζαν. Ο συλλαφισμός στην Ευρώπη προχωράει. Έχει καταγγελθεί από πολλούς και από το Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Ινάνς, ε, του Βελγικού κράτους, της Οργάνωσης για την Εκπαίδευση και από άλλους. Ισχύει στο Βέλγιο, στις κατοχώρες και αλλού ο σελαφισμός βρίσκεται πίσω από τους 800 ή 1000 που έφυγαν από την Ευρώπη θελοντές για να πάνε να πολεμήσουν με τους αντάρτες στη Συρία. Έχουμε απέναντί μας μια μεγάλη απειλή που προχωράει. Δεν λέω ότι είναι γιγάντια, δεν λέω ότι ο καθένας κρύβει έναν σελαφιστή, αλλά το να διαχωριστούν οι μουσουλμάνοι από τους μη μουσουλμάνους με προκλήσεις είναι ένα καθημερινό φαινόμενο και η τρομοκρατία των σαλαφιστών είναι κάτι που το έχουμε δει τους τελευταίους 12 μήνες. Από το 2005 μέχρι το 2012 στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπήρξε καμία επιτυχής επίθεση, ενώ τους 12 τελευταίους μήνες είδαμε. Υπάρχει επέκταση δηλαδή του κινήματος. Για το Σουρασέρ δεν χρειάζεται. Να επανέλθω νομίζω ότι απάντησε ο συνάδελφος. Είναι σαφές ότι αν οι σελαφιστές χάσουν στη Συρία θα υποχωρήσουν. Αλλά και πάλι σας παραπέμπω σε αυτά που είπε ο κύριος Σαριμόρα. Οι σχέσεις σελαφιστών και ουχαμπιτών που με ρωτήσατε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία διάρθρωση δύσκολο να την καταλάβει κανείς. Χοντρικά, οι οχαμπιτές ασχολούνται πιο πολύ με το θέμα του κύριου Ρασιμόρα, δηλαδή με την προπαγάνδα. Με το ψυχολογικό έργο, η διαπαιδαγώγηση αν θέλετε. Και δεν δρούν τόσο πολύ, ενώ οι σαλαφιστές έχουν επωφεληθεί από χρηματοδότηση ακόμα και των ουαχαμπιτών για τις δράσεις τους. Τέλος, για την Σαουδική Αραβία. Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει χρηματοδότηση που κατέληξε σε τρομοκρατικές οργανώσεις και Αλκαΐντα και άλλες από τη Σαουδική Αραβία. Μερικές φορές μάλιστα από άτομα πολύ ψηλά στην κοινωνική κλίμακα, ακόμα και από την ε, άρχουσα τάξη και τη βασιλική οικογένεια. Σήμερα έχουμε συνεργασία, ειδικέ υπηρεσίες της Οδικής Αραβίας και της Αμερικής, αρκετά ικανοποιητική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αλλά από ιδιώτες εξακολουθούν να πηγαίνουν χρήματα από τη Σαουδική Αραβία στην τρομοκρατία. Η συνεργασία πάντω Οδική Αραβία, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπη είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο σήμερα για την καταπολέμηση πάντα τη τρομοκρατία. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Τέλο, συνάδελφοι, να σα υπενθυμίσω ότι το επόμενο θέμα είναι και κλεισμένο των θυρών, που σημαίνει ότι παρακαλώ όσοι δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην αίθουσα ή ε, δυνατόν να ε, βγουν και σε λίγα μόνο λεπτά θα ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα.